Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα εδώ. Καλώς ορίσατε στην δημόσια κρόαση που οργανώνει η Επιτροπή των Γυναικών προετοιμάζοντας την έκθεση για την ε. κατάσταση των γυναικών στην Βόρεια Αφρική. Όπως γνωρίζετε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων αποφάσισε να αφιερώσει ένα σημαντικό τμήμα της εργασία των εργασιών της φέτος σε αυτό το θέμα. Ξεκινάμε σήμερα με τη δημόσια κρόαση, μετά από την οποία η κυρία Κώστα η εξότιμη συνάδελφος θα συντάξει σχετική έκθεση. Και μετά μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας θα επισκεφθεί την Ισία στα τέλη του Οκτωβρίου. Ε, όλοι συμφωνούμε και αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο των γυναικών στην ε, αποκαλούμενη Αραβική Άνοιξη. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος πως οι δημογραφικές αλλαγές θα μπορούσαν ε, να επηρεάσουν δραματικά τη ε, δικαιώματα των γυναικών και ανησυχούμε πολύ γι' αυτό. Οι δημοκρατικές αλλαγές θα επηρεάσουν την κατάσταση των γυναικών. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε, ε, να δούμε ε, κατά πόσο έχουν δίκιο αυτοί που ονομάζουν αραβικό φθινόπερο την Αραβική Άνοιξη όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Πρώτη, η κύρια ερώτησή μας θα πρέπει να είναι τι, και τώρα τι γίνεται. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως οι γυναίκες δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τις αλλαγές για, και ότι θα ισχυ... δεν θα... και ότι η δημοκρατία θα είναι γνήσια και θα περιλαμβάνει και το γυναικείο ημίση του, του... του πληθυσμού. Οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ένα ε, δραστήριο ρόλο και να οθήσουν τις αλλαγές. Η συντάκτρια της νομοδότηση που ήδη έχει γίνει, η, κυρία Κορίνα Κρετού από τους σοσιαλιστές ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, αλλά έχουμε εμείς εδώ τη συντάκτριά μας, την κυρία Κώστα, στην οποία και θα δώσω αμέσω το λόγο. Εγώ θα μιλήσω Ιταλικά. Μάλιστα, κατα... Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Ειδίθ Μπάουερ που είχε την ευγενή καλοσύνη να οργανώσει αυτή την σημαντικότατη ακρόαση. Βλέπω εδώ και άλλους συνεδέλφους, την κυρία Ρομέρο και άλλους φαντάζομαι που θα έρθουν στη συνέχεια. Και είμαι πεπισμένη ότι η συνάντηση αυτή δεν θα είναι η τελευταία μας, διότι ως εισηγήτρια θα ήθελα να επιμείνω να γίνουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις τους επόμενους μήνες και επαφέ μέσω των δικτύων ή άλλων μορφών συνεργασίας. Πιστεύω. Ως γυναίκα δε και ως ευρωβουλευτής απο έρχομαι από μια χώρα όπως η Ιταλία που έχει βαθιές ιστορικές σχέσεις με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και ιδιαίτερα με τις τέσσερις χώρες που αντιπροσωπεύονται σήμερα εδώ, την Ισία, Αίγυπτος, Λιβύη και Μαρόκο, πιστεύω πως θα έπρεπε θα, έπρεπε καταρχήν να πω πως η σημασία, όπως έλεγε και η Edith Bauer, ως Επιτροπή Γυναικών μπορέσαμε να, συγκεντρώ, να, συγκαλέσουμε αυτήν την ακρόαση και να τη χρησιμοποιήσουμε και ως τρόπο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας για τις γυναίκες που ήταν η ε, πρωταγωνίστριες στα μεγάλα λαϊκά κινήματα που οδήγησαν στην Αραβική Άνοιξη και που σήμερα ε, με ελπίδες βλέπουν το μέλλον, αν και με κάποιες ανησυχίες, αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις ε, στην ε, χώρα σας. Και θα ήθελα να ακούσω από σας, ε, γιατί έχουμε εκπροσώπους πολύ σημαντικούς, ειδικέ δημοσιογράφους, υπεύθυνε ομοσπονδιών, ενώσεων και ΜΚΟ, εκπρόσωπους θεσμικών οργάνων, εν πάση περιπτώσει γυναίκες που μπορούν να δώσουν μια μεγάλη συμβολή ώστε να αρθεί αυτό το βέλο το οποίο καλύπτει τις δραστηριότητες από ε, τότε που άναψε αυτό το πρώτο λαμπύρισμα για αυτών των μεγάλων αλλαγών που έγιναν και πολύ συχνά οι νέοι και οι γυναίκες ήταν στην πρώτη γραμμή και δεν πρέπει να ξεχαστούν σήμερα. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο κάτι ακόμα ότι δηλαδή δεν μπορώ και πιστεύω και μιλώ και εξ ονόματος των άλλων συναδέλφων δεν μπορώ να σιωπήσω για τη σοβαρή κατάσταση που ε, σοβεί αυτή τη στιγμή στη Συρία που πιστεύω όλοι μας θα πρέπει να είμαστε πιο στεναροί στην καταγγελία και στις ε, αντίστοιχες δράσεις γιατί η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παρακολουθεί τις φαγές όπως την τελευταία της Χούλα που ε, έπληξε κυρίως γυναίκες και παιδιά είναι ένας λαός που δοκιμάζεται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξή στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω όθησης του Κοινοβουλίου ανέλαβε την ευθύνη, τη δεσμευσή να ενισχύσει την ευρωμασογειακή εταιρική σχέση ώστε να επανδύσει στις νέες ε, ε, δημοκρατίες σας με προγράμματα συνεργασίας στο ε, ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της, κοινωνικής, της κοινωνίας των πολιτών μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών εξελίξεων. Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ και το έχουμε δει σε πολλές άλλες ε, συγκρουσιακές καταστάσεις και μετά από αυτές ότι χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών, δηλαδή η συμμετοχή τους από κάτω, ε, από τη βάση ε, στους θεσμούς, η αναγνώριση του ρόλου των γυναικών και των δικαιωμάτων τους ως αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα οδηγήσουν ούτε σε δημοκρατή ούτε σε πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη. Και από αυτή την πεποίθηση ξεκινά ε, πηγάζει η βούληση αυτής της ε, Επιτροπής μας να συσφίξουμε τις σχέσεις, να συντάξουμε αυτή την έκθεση μαζί με τους ε, για να δώσουμε περισσότερη ισχύ σε αυτή την πεποίθηση. Είναι σημαντικό ότι νέα αυτή η πολιτική γετνίαση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2011 ορίζει μια νέα προσέγγιση επί τη βάση τεσσάρων βασικών αρχών. Η πρώτη είναι το more for more, περισσότερα για περισσότερα, περισσότερη στήριξη στις χώρες που θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη δημοκρατική μετάβαση. Αυτή είναι μια προσόγγιση που ε, ε, μολύνει, ας πούμε, μάλλον επηρεάζει και τις άλλες επιτροπές. Όπως... Χωρίς να τα μολύνει όμως. Και μια δεύτερη αρχή τώρα είναι η αμοιβαία υπευθύνη, υπευθυνότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιούχων. Αυτό μας οδηγεί σε μεγαλύτερη εταιρικότητα και ισότητα. Τρίτη, αρχή. Όχι μόνο να εμπλεκόμαστε σε, θετικό, σε θεσμικό επίπεδο, αλλά επίσης και το επίπεδο της κοινωνία των πολιτών, συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους τέτοιου φόρου. Θεωρείται αυτή τη σημαντική αρχή. Εκπεφρασμένη αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα μέσα στα πλαίσια της νέας αυτής εταιρική πολιτική, Ακόμα και στην πρώτη ανακοίνωση τη Κομισιόν που ανέφερε η ύπατος εκπρόσωπος για τα θέματα εξωτερικών πολιτικών της Κομισιόν στην πρώτη και στην πρώτη κοινή ανακοίνωση ήδη είχε προκαταλάβει τη σημασία των γυναικών στην πολιτική γειτονία. Και επίσης στο χώρο, ιδίως ιδιαίτερα στο χώρο της Μεσογείου. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας ειδικό εισηγητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωμεσογειακή περιοχή και ότι έχει δημιουργηθεί και μια σειρά από μονάδες κρούσης διμερούς επίπεδου. Η πρώτη θα είναι στην Τινησία και η επόμενη στην Αίγυπτο μετά τις εκλογές με στόχο τη δημιουργία συμφωνιών που θέτουν σε διάθεση των χωρών αυτών τους επαγγελματικούς, οικονομικούς και πολιτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένω είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς και πού οι γυναίκες της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρική. θα συνεχίσουν να εμπλέκονται σε συνεργασία στο μεσογειακό χώρο μετά από την πτώση των δικτατορικών καθεστώτων που για πάρα πολλά χρόνια είχαν παραμείνει αμετακίνητα, έχει δημιουργηθεί μια νέα δυναμική. Και επίση στα πλαίσια του Συμβουλίου τη Ευρώπη αρχίζουν να, εγκρίνονται διμερεί πρωτόκολλα συμμετοχή την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο με το Μαρόκο. Και επίση έχει γίνει δεκτή η νομοθετική πρόταση για το επόμενο εργαλείο γειτονία που θα λέγεται European Neighborhood Instrument. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα νέα εργαλεία τα οποία θα σύμβαση για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μια καλύτερη σχέση με τι χώρε αυτέ τη Βόρεια Αφρική μέσα στα πλαίσια τη υποστήριξη του ρόλου των γυναικών στι χώρε αυτέ. Ναι. Προβλέπετε λοιπόν να υπάρξει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκά, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 1 δισεκατομμύριο ευρώ και άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί με στόχο να μπορούμε να παρεύουμε με ταχύτητα για να υποστηρίξουμε την μεταδοτική μετάβαση, την ε, δημοκρατική συγγνώμη, μετάβαση με ειδικά εργαλεία. Επίση υπάρχει και ένα ειδικό εργαλείο που υποστηρίζει τι μη κυβερνητικέ οργανώσει τη χώρα αυτέ και την κοινωνία των πολιτών στου χώρου αυτού. Επομένω, μέσα σε αυτόν τον ευρύ ορίζοντα θα ήθελα και εγώ να τονίσω ποια είναι η δική μου θέση υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται η συνάντησή μα, Υπάρχει η σημαντική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα πρέπει να επενδυθεί πλήρω στη δυνατότητα να συμμετάσχει πλήρω στη δυναμική η οποία ανοίγεται σήμερα ενώπιόν μα και πιστεύουμε τον τρόπο αυτό έχουμε μια μείζωνα δυνατότητα συνεργασία σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο μεταξύ των εδώ γυναικών και των εκεί γυναικών από την άλλη οφθή τη Μεσογείου, διότι με τον τρόπο αυτό, όπω φάνηκε και από την γνωμοδότηση τη κυρία Μποσκούρτ, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι απαραίτητο να μιλήσουμε και για τη γυναικεία διάσταση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Εκεί εγγραφόμεθα. Ω εισηγήτρια, λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζω ποιε είναι οι δικέ σα προτάσει και δικέ σα αναλύσει για να καταλάβω καλύτερα την κατάσταση των γυναικών σε διάφορα πλαίσια. Γνωρίζω ότι οι χώρε σα είναι πολυπίκυλε ιστορικά, πολιτικά, πολιτιστικά, θεσμικά και συνταγματικά. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία έχουν εγκαρσιότητα και οριζοντιότητα σε όλε αυτέ τι χώρε τη Βόρεια Αφρική σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και την νέα εμπειρία από την Αραβική Άνοιξη. Πιστεύω λοιπόν μετά από όλα αυτά ότι θα πρέπει επίση να επιζητήσουμε βάσει των ενδείξεων που θα μα δώσετε πώ θα μπορέσουμε να έχουμε τι δικέ μα θέσει. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη μα στις προσπάθειες που καταβάλουν για την ευρωπαϊκή πολιτική μεσογειακής γειτονίας, ώστε να έχουμε σταθερές σχέσεις μέσω και των διμερών αντιπροσωπείων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Κοινοβουλίων των χωρών σας, οι οποίες είναι εν εκτιδίξη και μετά από όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά στο σεβασμό Τη αυτονομία και των επιλογών, πολιτικών και θεσμικών επιλογών που είναι αυτόνομες για τις χώρες, αυτό, αυτές δηλαδή στις οποίες προβαίνεται, καθώς και τον πλουραλισμό τον θρησκευτικό που εκφράζεται και ως γυναίκες και νομίζω πως θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο προβοκύπτει από, από τόσες ε, διεθνείς συμβάσεις σκέφτομαι το Πεκίνο, τη ΣΥΝΤΟΒ, την Διεθνή Σύμβαση κατά των διακρίσεων θα πρέπει λοιπόν να θα ήταν χρήσιμος ένας διάλογος και μια αντιπαράθεση ώστε να μιλήσουμε για τις καθολικές mm. αρχές ε, για τον άνθρωπο, για τη γυναίκα και τον άνδρα, ισότητα και ισότητα δικαιωμάτων. Θα πρέπει να σας πω από προσωπική εμπειρία πως δεν είναι μόνο δυνατόν αλλά είναι απόλυτα συνεπές το να συνδυαστεί η πίστη, η θρησκευτική πίστη με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ε, αδέλφια ενός μόνου πατέρα. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να βελτιώσουμε τη βάση της αμοιβαίας συνεννόησης και συνεργασίας. Πέρα από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που κάποιες φορές ισχύουν και για τις γυναίκες. Θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα το εξής. Όπως ε, αυτές τις μέρες μας φαίνεται, γιατί ξέρουμε και πω αυτές τις μέρες γίνεται μια ε, διαδήλωση στην πλατεία Ταχρήρ κατά το, της έκβασης των τελευταίων προεδρικών εκλογών, κατά της βίας. Να ξέρουμε αν αυτές οι δημοκρατικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν, αν εκεί οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται και αν προωθούνται τα δικαιώματά τους και κυρίως αν αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό που να σέβεται τις προσδοκίες των γυναικών και των νέων, αλλά όχι μόνο σκέφτομαι τις διαφορές, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορές τεράστιες ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο και σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών και τις απαιτήσει τους, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για κάποια στάδια τα οποία ήταν σημαντικά, αλλά και που θα μπορούσαν ε, επίσης να είναι αντιφατικές αυτά τα στάδια. Πρώτο θέμα λοιπόν φέτος είναι η μεγάλη συμμετοχή των γυναικών, όπως είπαμε, στις πρώτες ελεύθερες ε, και δημοκρατικές εκλογέ ήταν για πολύ μεγάλη. Ε, Περνάμε λοιπόν από 27% των γυναικών βουλευτών στην Τινησία παρότι δεν έγινε σεβαστή η ποσόστοση αλλά μόνο μια ένδειξη εναλλαγής ανάμεσα σε άνδρες ε, και γυναίκες περνάμε στις τρεις γυναίκες υπουργού φέτος από το 3% χάρη στις ποσοστώσεις με μια γυναίκα υπουργό μέχρι το 2% της Αιγύπτου με μόνο δύο γυναίκες στην κυβέρνηση αλλά και λόγω του αποκλεισμού τους από την πολιτική μετάβαση παρά το ότι η blogger Ασμάου είχε, είχε ξεκινήσει την πρόσκληση για διαδήλωση στην πλατεία Ταχρή τον Ιανουάριο του 2011 και μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ φέτος. Ε, Σκέφτομαι επίσης το 5% των ε, Λίβιων γυναικών με δύο γυναίκες ε, στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στο πριν και το μετά και δεν μετριέται μόνο με τα, τους αριθμούς. Αυτή τη στιγμή Έχουμε όντω ελεύθερε και δημοκρατικές εκλογές και είναι διαφορετική η εκπροσώπηση των γυναικών που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο από, ε, πριν, από ότι πριν όπου ορίζονταν γυναίκες ε, από, εκ των άνω. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε αν υπάρχει αυτή η αίσθηση αυτό που διαβάζουμε σε πολλά σχόλια και στον τύπο και στον τοπικό σας ε, τύπο, ότι γενικά γίνεται μια απόπειρα να περιθωριοποιηθούν σε αυτή τη φάση οι γυναίκες και οι νέοι μετά από την Επανάσταση και λόγω της νίκης ε, Ισλαμιστικών κομμάτων, αν και με διαφοροποιήσεις και διαφορετικούς συνασπισμούς, που είναι και, αυτοί πολύ ενδιαφέροντες, ή αν υπάρχει ευθύνη και λόγω του μεγάλου κατακαιρματισμού των, ε, εκλο... των ψηφοφόρων. και των κομμάτων που μπήκαν ας πούμε στον, στον αγώνα αλλά με διαφορετικούς ε, τρόπους και, και σχετικά με ελλειπή οργάνωση. Και για την Αίγυπτο κυρίως, ε, τι πιστεύετε ότι αυτή, τη στιγμή στην Αίγυπτο ε, Έχουμε δύο υποψηφίου που θα συμμετέχουν στην επόμενη, στις επόμενες εκλογές, ο Φίκα και Μόρση. Ο ένας, κατά κάποιο τρόπο, είναι στρατηγικός και κοντά στο καθεστώς της προηγούμενης κυβέρνησης και ο Μουρσί που είναι με ένα από τους αδερφούς μουσουλμάνους αλλά που προτείνει ένα, μια κυβέρνηση θρησκευτικού τύπου. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν ποιο είναι ο προσανατολισμός των γυναικών για αυτές τις επιλογές που είναι επιλογές οι οποίες είναι πολύ αντιφατικέ. Δεύτερο ε, ερώτημα. Η συντακτική διαδικασία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Στην Αίγυπτο ενεκρίθη μια πρώτη μεταρρύθμιση με ένα δημοψήφισμα το 2011, αλλά η πραγματικό σύνταγμα θα εγκριθεί από μια επιτροπή που θα οριστεί από το ίδιο το Κοινοβούλιο μετά από τι προεδρικέ εκλογέ και σκέφτομαι και τη συντακτική συνέλευση όπου οι γυναίκες είναι το 27% των βουλευτών στην Τινησία και εκεί θα εγκριθεί το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα που ήδη εγκρίθηκε στο Μαρόκο, ενώ στη Λιβύη εγκρίθηκε ένα σύνταγμα για τη μεταβατική περίοδο μέσα στη διάρκεια του 2011. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτά τα συντάγματα υπάρχει γενικά μια αναφορά πολύ ρητή στο θέμα της ισότητας, ε, στην κατάργηση των ε, διακρίσεων, βέβαια με διαφορετική νομική ισχύ. Ε, ξέρω πως οι γυναίκες θέλουν να θεσμοθετήσουν το δικαίωμα της ισότητας κτλ. Αλλά στην Ισία που νίκησε ένα μετριοπαθές Ισλαμιστικό κόμμα το Εναντά, το οποίο δεν αναφέρει στο κείμενο την Σαρία, ακόμα και αν η μουσουλμανική θρησκεία είναι η κύρια στην Ισία. Ε, αυτό είναι ε, περισσότερο αδύναμο από ό,τι στο Σύνταγμα του Μαρόκου, της Λιβύης και της ε, Αιγύπτου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση στα συντάγματα, αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πολλές επίσημες δηλώσεις αυτών των κυβερνήσεων και των κομμάτων ήταν σημαντικές γιατί είπαν ότι η ισότητα θα είναι εγγυημένη, ότι θα ισχύσει η αρχή των μη διακρίσεων, ότι θα καταργηθούν τα αποθέματα για ε, τα, οι, συγγνώμη, επιφυλάξεις για τη σύμβαση ΣΥΝΤΟΥ και μιλώ για την Ισία, αλλά και στην Αίγυπτο είπε τα ίδια η κυβέρνηση αν και ακόμα δεν προέβησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Αλλά ενώ το λένε αυτό, υπάρχουν και ανησυχητικές δηλώσεις. Ε, πιστεύω πως στην Ισία, ας πούμε, κάποιοι πολιτικοί μίλησαν κατά των υιοθετήσεων, κατά των... Ε, ε, ανήπαντρων μητέρων Είπαν επίσης ότι δεν θα προχωρούσαν στον ορισμό γυναικών ως δημάρχων. Ε, υπάρχουν δηλαδή κάποιες πρόοδοι, αλλά ενώ ταυτάχρονα ε, ε συνεχίζουν να υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, ε, οπισθοδρομικές ε, καταστάσεις και επίσης η σχέση των ΜΚΟ ήταν πολύ σημαντική γιατί αυτή η συμμετοχή χρειάστηκε να ενισχυθεί ας πούμε τρεις ΜΚΟ στο Μαρόκο έδωσαν ε, την θέση τους σε ένα συνασπισμό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Γυναίκες στις Γυναίκες το οποίο φέτος ε, ορίστηκε εκ νέου. Υπάρχει διαφορετικό είδος συμβουλίου, αλλά με ποιο τρόπο θα συμμετέχει, θα ήθελα να το καταλάβω. Και επίσης, ποιος είναι ο τρόπος, ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν οι, οι, οι πώς συμμετέχουν στην εθνική πολιτική. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πως ε, ο ρόλος των ΜΚΟ με τη μορφή της συνεργασίας ε, και της ε, ανάπτυξης εντείνεται. τώρα, η διαφορά της θέσης των γυναικών μεταξύ των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Περνάμε από το 75% των εκπαιδευμένων γυναικών, ένα πολύ ψηλό επίπεδο στην Τινησία, και σε σχέση με τις ε, προγραμμα... προγραμματικές δηλώσεις των κυβερνήσεων. Ποιες είναι οι προτεραιότητες επί των οποίων γίνονται επενδύσεις ε, και πού μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις Ευρωπαίες γυναίκες και τις γυναίκες ε, της Βορειοαφρικής. Ας πούμε, πρόσβαση στο υγειονομικό σύστημα, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην πίστοση. Ε, ε, έτσι ώστε να φτιάξουμε κατά κάποιο τρόπο ε, μια ατζέντα ευρωμεσογειακή. Έχουμε τώρα το θέμα των ΜΜΕ. Έχουμε εδώ μια εκπρόσωπο δημοσιογράφο ένα στοιχείο. Τις προάλλες ορίστηκαν τρεις γυναίκες επικεφαλής τριών κρατικών ραδιοφωνικών σταθμών στη Ισία. Ένα πολύ θετικό στοιχείο ε, σε άλλες περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν μπει λίγο στο περιθώριο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας σε άλλες χώρες. Σε σχέση με όλα αυτά, ο ρόλος των ΜΜΕ, των ανεξαρτήτων και των γυναικών σε αυτά, θα θέλαμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς προχωράνε τα πράγματα. Και έπειτα ακόμα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την νομοθεσία. Τις νομοθεσίες στις χώρες αυτές που εξακολουθούν να ε, καθιερών ε, διακρίσεις θα μας το πει αυτά η συνάδελφος από τη Λιβύα που είναι πολύ ειδική όσον αφορά τα θέματα για τις βίες και τις βίες κατά των γυναικών ξέρουμε πως χρησιμοποιήθηκε ως όπλο και κατά τη διάρκεια της ε, επανάστασης για να εκφοβιστούν οι διαδηλωτές αλλά ξέρουμε και το εμπόριο γυναικών ε, ανθρωπίνων όντων η συνάδελφος Ρομέρο έχει ασχοληθεί πολύ και η συνάδελφος Μπάουερ που ήταν συγγήτρια για την εμπορία των ανθρωπίνων όντων ε, συμμετείχε ε, ενεργά και ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό ότι δυστυχώς σε χώρες όπως η Λιβύη συχνά η εμπορία σημαίνει άλλες Αφρικανές γυναίκες, μετανάστριες. Η Λιβύη συχνά είναι χώρος διέλευσης, γίνεται πολύ μεγάλο εμπόριο. Πριν, το είχαμε αυτό πει πριν από τρία χρόνια, πριν να γίνει η Επανάσταση και θα θέλαμε να φτιαχτεί μια πραγματική συμμαχία ανάμεσα στις γυναίκες του Ευρωκοινοβουλίου και τι γυναίκες αυτών των χωρών για να αποφύγουμε τέτοιες μορφές ε, σοβαρότητα τη εκμετάλλευσης που αποτελούν στην ουσία την ε, ε, δουλεία αυτού του αιώνα. Εγώ λοιπόν σας, ε, έδειξα, σας είπα κάποια θέματα στα οποία θα μπορούσατε να μας πείτε τις απόψεις σας. Ε, έχουμε μια ευκαιρία σήμερα πολύτιμη για να αναλύσουμε τα θέματα και για να ακούσουμε τις δικές σας κρίσεις, αντιδράσεις και τις δικές σας προτάσεις σε σχέση με τις δράσεις που θα μπορούσαμε από κοινού να κάνουμε. Για την έκθεση προβλέπετε τον Ιούλιο να έχουμε μια, μάλλον τον Οκτώβριο θα, υπο, θα παρουσιάσω την έκθεσή μου, μετά θα υποβληθούν οι τροπολογίες και σε εκείνη την περίοδο, νομίζω στα τέλη του Οκτωβρίου θα κάνουμε μια επίσκεψη στην ε, στην Τίνιδα θα είναι μια ευκαιρία για να σας ακούσουμε ακόμα μια φορά και μετά στη συνέχεια θα εγκριθεί η, η, έκθεση και έχουμε μισά για άλλη μια ακρόαση μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά για να σας πω ότι πραγματικά ελπίζω πως ξεκινά μια νέα εποχή στις σχέσεις μας και είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να συμμετέχω μαζί με τις υπόλοιπες συναδέλφους. Ευχαριστώ. Thank you so much, Σας ευχαριστώ πολύ Σιλβία που χρησιμοποίησατε με φιδό το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Θα ήθελα τώρα να χαιρετήσω τις διακεκριμένες ομιλήτριές μας και να τους δώσω το λόγο. Όπως βλέπετε έχουμε ένα μακρό κατάλογο ερωτήσεων, δεν έχουμε πολλές απαντήσεις. Η ελπίδα μου είναι ότι στο τέλος της ημέρας και της ακρόασης η κατάσταση θα είναι λίγο πιο σαφής. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στις δύο πρώτες διακεκριμένες ομιλήτριές μας την κυρία Σόντεσμεν Χαλίφα από την Τινησία. Είναι δημοσιογράφος στο ε, ραδιόφωνο της Διεθνούς ε, Αλυσίδας, την Asian Chain International και έχει συμμετάξει σε πολλές διασκέψεις για το ρόλο των γυναικών στα μίδια και ασχολείται με το θέμα με το πώς οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ένα οδηγό ρόλο στην αλλαγή στη Βόρεια Αφρική. Η δεύτερη ομιλήτριά μας η κυρία Στουάτ Βέιντι, πανεπιστημιακή και εκπρόσωπος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα δικαιώματα γυναικών από τη Λιβύη. Η κυρία Βέιντι είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, ενεργό μέλος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που έχει σε στόχο την προώθηση των γυναικών σε αγροτικές περιοχές της Λιβύης και από το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους εμπλέκεται στην προστασία γυναικών που έχουν τύχει θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια της καταστολής μετά την Αραβική Άνοιξη. Ήταν προηγουμένω εμπειρογνώμων για τα θέματα φύλου του Μεταβατικού Συμβουλίου, υπουργό Γυναικείων Θεμάτων και έχει δημιουργήσει πρόσφατα μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει σαν στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών Κυρία Σόντες θα σας δίνω το λόγο λοιπόν. Θα Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου ενώπιόν σας. Θα αρχίσω με ένα ιστορικό της εξέλιξης του θέση της γυναίκας στην Τινησία, γιατί θεωρώ ότι χωρίς μέλλον δεν υπάρχει ούτε παρόν ούτε τίποτα. Χωρίς παρελθόν, μα χωρίς τη γνώση του παρελθόντος δεν υπάρχει μέλλον, ούτε και παρών. Η ισότητα των φίλων στην Τινησία προκύπτει από την ομοθεσία αλλά έχει εξελιχθεί μέσα στο χρόνο το οικογενειακό δίκαιο και ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία έχουν αλλάξει πολύ. Στην Τινησία μπορεί κανείς να πει ότι για πολύ καιρό υπήρξε μία πρωτόγνωρη εμπειρία στον αραβικό κόσμο ως προς τις γυναίκες. Το Σύνταγμα της Τινησίας κατήργησε την πολυγαμία, εγκαθίδρυσε την νομική ισότητα ανδρών και γυναικών αγάμων και εγγάμων και αυτό έδωσε στις γυναίκες ε, μια νέα έννοια της ελευθερίας και του χαρακτήρα τους ως πολιτών. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρξε στις άλλες χώρες του αραβικού κόσμου. Έχουν δικαίωμα στην έκτρωση, υπάρχει ένα εγγυημένο ποσό στην περίπτωση που η γυναίκα υπανδρευθεί και συνέχισαν, συνεχώς ζητούσαν περισσότερα δικαιώματα ακόμη και υπό τον Μπεναλή σε θέματα διαζυγίου και ηθαγενείας καθώς και καταπολέμησης της οικογενειακής βίας έκαναν μεγάλες πρόοδους οι γυναίκες γιατί τιμωρείται η οικογενειακή βία. Υπό το καθεστώς του Μπεναλή έδωσαν έναν τελευταίο αγώνα για το κληρονομικό δίκαιο. Εκτός αν υπάρχουν προβλέψεις των γονέων τους, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα σε πλήρη κληρονομία και περιορίζεται επομένως ακόμη και σήμερα ο ρόλος του στο ρόλο της ε, τεκνοποιίας. Καταλαβαίνετε όμως γιατί το καθεστώς του Μπεναλή έλεγε ότι είναι φραγμός κατά των Ισλαμιστών. Το προηγούμενο λοιπόν αυτό καθεστώς κατεμένα έδινε στις γυναίκες το ρόλο, δευτε, ε, δευτερεύοντα ρόλο στην πολιτική σκηνή. Και γι' αυτό οι γυναίκες κατέληξαν να γίνουν ο ακρηγωνιαίος λίθος της Επανάστασης γιατί ήταν οι πρώτες που κινητοποιήθηκαν από το 10 ήδη και οι εξελίξεις οδήγησαν στην πτώση του Μπεναλή. Άνδρες και γυναίκες ε, έπαιξαν ισότιμο ρόλο στην καταπολέμηση της δικουτατορίας. Σήμερα το πρόβλημα είναι άλλο. Η Επανάσταση βελτιώνει τη θέση των γυναικών. Μετά τις 14 Ιανουαρίου είδαμε αντιφατικές εξελίξεις στην Τινησία ως προς τις γυναίκες. Οι πολιτικοί πρωταγωνιστές είπαν αντιφατικά πράγματα. Η χώρα πάντως μπορεί να περηφανεύεται ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία του αραβικού κόσμου. Γιατί είναι υποχρεωτικό να σέβονται όλη την ισότητα των δύο φύλων και στις εκλογές, ε, δεν φάνηκε αυτό. Υπήρξε μεγάλη παρουσία γυναικών στην πολιτική ζωή, απ' την άλλη όμως η μεταβατική κυβέρνηση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αποτελείται από άντρες. Λιγότερο από 20% γυναικών συμμετείχαν στη μεταβατική αυτή κυβέρνηση και οι εκλογικές αρχές στις εκλογικές αρχές μόνο δύο γυναίκες στα 16 μέλη παρατηρήθηκαν. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη ανισότητες και αυτές Τις καταδικάζει το φεμινιστικό κίνημα που δυστυχώς αντι... στο οποίο δυστυχώς αντιδρούν οι συντηρητικές δυνάμεις και θέλουν μείωση του ρόλου των γυναικών στην επαγγελματική ζωή. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για τις γυναίκες και οφείλεται εξ ολοκλήρου στο συντηρητισμό. Δεν θέλουν πάντως να εγκαταλείψουν τα κεκτημένα τους η Τρόικα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία λέει ανεπίσημα ότι δεν θα θίξει το οικογενειακό καθεστώς ή το καθεστώς των γυναικών και γι' αυτό συνεχίζουν τον αγώνα τους οι γυναίκες και για τη δημοκρατία και για την ταυτότητα. Είναι στην πρωτοπορία για την καταπολέμηση του φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας για την ανεξιθρησκεία και για την ισότητα των φύλων. Κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις, συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί τάσσονται στεναρά υπέρ της ισότητας των φύλων και του μοντερνισμού. Βέβαια μεγάλο μέρος του πληθυσμού πιστεύει ακόμη τα σκοτα... τη σκοταδιστική προπαγάνδα. Ορισμένοι σαλαφιστέ και σαλαφίστριες που δεν παίζουν άλλο ρόλο εκτός από θρησκευτικό έχουν αυτές τις συντηρητικέ απόψεις αλλά αφού δεν παίζουν πολιτικό ρόλο δεν μας πειράζει αυτό. Το Εναχντά πάντως έχει υποσχεθεί να σεβαστεί το, τα δικαιώματα και υπάρχουν παρόλα αυτά άλλα κόμματα, μικρά κόμματα ισλαμιστικά που ζητούν την υποχρεωτική υποχρεωτικά τον Φερετζέ και ε, ιδίως το κόμμα Ταχρέρ όχι το Εναχντά που είναι στην εξουσία οι περισσότερες γυναίκες θεωρούν ότι η νίκη των Ισλαμιστών του Εναχντά θα βλάψει τα δικαιώματά τους, θα τις ζημιώσει αλλά αυτό εξαρτάται από την πολιτική θέληση που θα επιδείξει η κυβέρνηση αυτή αν θέλει όντως να προστατεύσει αυτά τα δικαιώματα. Πρέπει να ελπίζουμε ότι η κοινωνία των πολιτών και η δημοκρατική κοινωνία γενικότερα θα δώσει στις γυναίκες το ρόλο που τους αρμόζει. Βρισκόμαστε σε καμπή διότι τώρα συγγράφεται το σύνταγμα, το καινούργιο σύνταγμα και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει η ισότητα των φύλων να εμφαίνεται εκεί ως βασική αρχή απαράβατη. Δεύτερον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα και ιδιαίτερα τα γυναικεία. Από το 59 είχε πει η Τινησία ότι οι διεθνείς συνθήκες θα γίνονται σεβαστές πέραν του εθνικού δικαίου και από αυτού δεν πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση. Ο αγώνας για την ισότητα των φίλων δεν θα είναι εύκολος και αν χάσουμε τον αγώνα αυτόν, αυτό δεν θα οφείλεται στο, σε κανένα κόμμα, ούτε αυτό που είναι στην εξουσία, ούτε στα Ισλαμιστικά, αλλά θα φταίνουν οι ίδιες οι γυναίκες. Θα ήθελα τώρα να σας πω, δείξω μερικές εικόνες από την ζωή των την ισίων γυναικών από την ανεξαρτησία. Εδώ μια αγωνίστρια εδώ βλέπετε μια αγωνίστρια. Για να δω. Μια αγωνίστρια. Όχι, ε. όχι αυτό είναι στην Επανάσταση. Παρακαλώ βάλτε το άλλο, την άλλη διαφάνεια πριν. Εδώ βλέπετε αμέσως μετά την ανεξαρτησία ότι βρίσκονται οι γυναίκες στο δρόμο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των. Μετά, μετά ε, θα έλεγα ότι ευτυχώς ο Χαντέ Μποργκέμπα τις υποστήριξε υποστήριξε εδώ είναι Φαχατεσέτ δεν βλέπω ακριβώς τι λέει αλλά Ναι, Τι υποστήριξαν και ο Μπουργκίμπα και ο Φερχάτα Σέτ. Τις υποστήριξαν. Ο Μπουργκίμπα και ο Φερχάτα Σέτ. Εδώ είναι η πρώτη γυναίκα ιατρός της Τινησίας. Εδώ είναι στην Επανάσταση. Ήμουν και εγώ εκεί. Ήμουν και εγώ εκεί. Επανάσταση. Υπάρχουν γυναίκες με φερετζέ, χωρίς φερετζέ, αγρότησες, πολίτησες και εδώ βλέπετε μία φοιτήτρια που σύει την σημαία, επισύει την σημαία Εδώ βλέπετε την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιείται. Όταν λέω δραστηριοποιείται, ναι μεν, αλλά όπως είπα και πριν και το ξαναλέω, μία κινητοποιούμενη κοινωνία των πολιτών κινητοποιείται καμιά φορά αρνητικά, δηλαδή απλώς αντιδράει και δεν δράει δεν έχει σαφή στρατηγική. Βγαίνουν στον δρόμο με πανό και τέτοια, αλλά, αλλά να. Αλλά. Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας αναφέρω, να σας δείξω και ένα βίντεο που με σημάδεψε. Το βρήκα κατά τύχη. Σημάδεψε. Να. Τον ήχο παρακαλώ. Δεν έχω ήχο. χωρίς μικρόφωνο. Α, εδώ δεν είχε ήχο, δεν ξέρω γιατί. Όταν το έβλεπα σπίτι μου είχε λοιπόν. Ε, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν ταξικές διαφορές και φιλετικές φίλων δηλαδή. Την νησία είναι την νησία όλων. Δεν υπάρχει χώρος για την ανεξιθρησκεία, την διακριτική μεταχείριση κτλ. Να, αυτό ήθελα να σας δείξω, δεν πειράζει που δεν είχε ήχο, τι να κάνουμε. Και άλλοι χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα να τελειώσω με μια θετική νότα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Τινησία και την Τινήσια. Να ξεπεράσει τον φόβο, δεν έχει φόβο, την ανησυχία γιατί όταν κανείς ανησυχεί δεν μπορεί να αντιδράσει <clears throat> όπως πρέπει. Πώς για τα μέσα ενημέρωση, ναι, ναι τα είπα και αυτά λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σουατουέιντι από τη Λιβύη στα ψηφοδέλτια, αυτοί ήταν πάντα άντρες. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η αριθμοί να είναι ισότιμοι, αλλά και στις εκλογικές περιφέρειες. Γενικά λοιπόν τα πολιτικά κόμματα δεν επέμειναν τόσο πολύ να είναι και γυναίκες ισότιμα πρώτες στο ψηφοδέλτιο. Παρόλα αυτά, από τις 27 έδρες στη Συντακτική Εθνοσυνέλευση από το σύνολο των εδρών μάλλον μόνο 59 είναι γυναίκες και οι περισσότερες από το ίδιο κόμμα βέβαια από το πρώτο κόμμα από το Εναχαντά Κάτι που παρατηρήσαμε στην έκθεσή μας ήταν ότι το σύστημα αυτό ισότιμης εκπροσώπησης θα μπορούσε να βελτιωθεί και στο μέλλον να περιλαμβάνει και ισότητα, ισότιμη εκπροσώπηση για τους πρώτους των ψηφοδελτίων. Uh, Κάτι άλλο σχετικά αρνητικό ήταν η κάλυψη από τον τύπο. Πολύ λιγότερο παρουσιάζονταν γυναίκες στον τύπο από κάθε κόμμα. Αυτά για τις εκλογές. Έπειτα Μετά τις εκλογές ακούστηκαν ανησυχίες ότι η συντακτική συνέλευση που γράφει το Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει πολλές γυναίκες, αυτό είναι ανησυχητικό. Αλλά επίσης το γεγονός ότι από αυτές τις γυναίκες 40 από τις 59 είναι από το μουσουλμανικό κόμμα Εναχδά. Εμένα αυτό με ανησυχεί γιατί η Εναχδά βασίζεται στο πρότυπο της Τουρκίας και τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε πολύ αρνητικά νέα από την Τουρκία ως προς τα δικαιώματα των γυναικών. Τίθενται λοιπόν ορισμένα απορίες και ερωτήματα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι μόλις έρχομαι από μια επιτροπή αυτού του συντονισμού της επιχείρησης των εκλογών που συζήτησε πώς θα μπορούσε το κοινοβούλιο μας να στηρίξει τα νεοεκλεγέντα μέλη της συντακτικής εκείνης εθνοσυνέλευσης, ας πούμε. Ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρατηρεί μαζί με τον ΟΗΕ την εφαρμογή ενός μεγάλου στηρικτικού προγράμματος για τα νέα μέλη της συνέλευσης που θα συμπεριλαμβάνει και υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών. Μερικοί από τα μέλη της συνέλευσης θα έρθουν και εδώ για να πάρουν πληροφορίες και ίσως αυτό να ήταν μια ευκαιρία να εκφράσουμε και εκεί σε εκείνους την υποστήριξή μας όλων αυτών που ανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Όχι, θέλω να κάνω κάτι διορθώσεις. Ήμουνα μέλος της εκλογικής επιτροπής που συνέταξε τον εκλογικό νόμο και ήθελα να κάνω διορθώσεις, αλλά τέλος πάντων. Μα ξέρετε, παρακαλώ κατανόηση ζητώ. Πρέπει να μιλήσει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η Μαρία Πιλάρ Πάμερο Μαλίγιο και κάποιος άλλος. Ποιος θα λάβει το λόγο πρώτος δεν το ξέρω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε τις ομιλήτριες γιατί και για μας είναι ευκαιρία να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Και για μας είναι σαφές και προτεραιότητα στα προγράμματά μας ότι σε συνεργασία με την Ευρωμέδ προετοιμάζουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Σεπτέμβριο 7 εκατομμυρίων ευρώ που θα ασχολείται ακριβώς με το θέμα της ισότητας των φύλων και για μας λοιπόν είναι προτεραιότητα όπως και η διαδικασία της Βαρκελόνης. Πάντοτε ανέκαθεν ήμασταν υπέρ της ισότητας των φύλων στην Βόρεια Αφρική δεν έχουμε τίποτε άλλο να προσθέσουμε. Να. Αν θέλουν να θέσουν τίποτε οι συμμετέχοντες, εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Σας κατευχαριστούμε. Έχουμε εδώ και άλλο πασκεκλημένο διακεκριμένο από τις εξωτερικές υπηρεσίες, την κυρία Γκλώριος Φερνάντες Κοτέρος Ακάδες. Μήπως θέλει να μιλήσει. Α, με συγχωρείτε, δεν λέγομαι Γκλώρια καταρχήν. Ήθελα απλώς να πω μερικά λόγια ότι και εμείς για να ακούσουμε ήρθαμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εμείς παίξαμε ρόλο και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την Επανάσταση. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τη διαφορά που έχει σημειωθεί στην Τινησία πριν και μετά την Επανάσταση, όπως είπε η μη κυβερνητική, η πρόσφαση της ΜΚΟ από την Λιβύη. Αλλά δεν ήταν ίδιες όλες οι επαναστάσεις. Θα επανέλθουμε μετά για το Μαρόκο, την Αίγυπτο κτλ. Αλλά εκεί θα φανεί ακόμη περισσότερο ότι δεν ήταν ίδιες οι επαναστάσεις. Εδώ θέλω να τονίσω ότι, όπως είπε και η κυρία Κώστα στην αρχή, το γενικό πλαίσιο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η πολιτική γειτονία. Αλλά και για την Τινησία και για το Μαρόκο και για άλλες χώρες έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίες σύνδεσης και σχέδιο δράσης πολύ προχωρημένο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα γυναικεία δικαιώματα. Τα έχουμε προετοιμάσει τα πράγματα. Και εγώ πήγα σε αντιπροσωπεία στην Τινησία, είδα την Επανάσταση εκεί και είναι ενδιαφέρον, όπως είπε η κυρία Χαλίφα, να μην ξεχνάμε το παρελθόν που υπάρχει εκεί. Ενώ με τη Λιβύη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί αρχίσαμε από το μηδέν και αρχίσαμε μερικά προγραμματούλια και προγραμματάκια για το εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να αρχίσει να γίνεται κάτι. Είναι η αρχή της αρχής για κάποια μελάχιστη διακυβέρνηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπέρ των γυναικών ενώ για την Τινησία τα πράγματα ήταν πολύ πιο προχωρημένα δεν υπάρχουν μόνο μικροπρογράμματα αλλά πραγματική βοήθεια και στήριξη για τον προϋπολογισμό, για την παιδεία, για την οικονομία, συγκεκριμένα προγράμματα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα στήριξη και υποβοήθηση mainstreaming που λέμε και στα γαλλικά. Εδώ πάντως ήρθαμε για να ακούσουμε. Σημειώνω μόνο ότι αρχίζει αμόλυση η διαδικασία αυτή. Από τώρα ως τον Οκτώβριο θα ακούσουμε ό,τι έχουμε να ακούσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προτού ξεκινήσω τώρα την ε, δεύτερη ομάδα των ομιλητών. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Βασίτ αν θέλει να απαντήσει σε αυτά τα οποία έλεγχαν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη χρήση του λόγου, απλώς για να δώσω ορισμένε πρόσθετες πληροφορίες Εμείς είμαστε μεταξύ αυτών που είχαμε προετοιμάσει την νομοθεσία για τις εκλογές. Στην Τινησία σε ό,τι αφορά το εκλογικό δίκαιο βρισκόμαστε σε παρθένο έδαφος γιατί ο νόμος που είχε ψηφιστεί ήταν ο νόμος για τις πρώτες εκλογές. <clears throat> Δεν θα ήταν ο οριστικός νόμος ο οποίος θα ίσχυε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πια καθόλου νομοθεσία. Δεν ξέρω αν το επόμενο σύνταγμα θα οδηγήσει σε ένα σύστημα εκλογών με απλή αναλογική ή πλειοψηφικό ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα είναι κοινοβουλευτικό το καθεστώς ή προεδρικό ή μη προεδρικό. Για τίποτα λοιπόν από όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βελτιώσουμε λοιπόν αυτό το σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν είναι η ύπαρξη πολλών πολιτικών κομμάτων που έκανε να εκπροσωπούν οι γυναίκες 23% από τους 217 που ήταν μέλη της συντακτικής συνέλευσης. Οι περισσότεροι εκλογικοί κατάλογοι ήταν με ανεξάρτητους ε, υποψηφίους. Υπήρχαν πάνω από 700 ανεξάρτητοι υποψήφοι. Γι' αυτό χρειάστηκε να ζητήσουμε μια ισότητα για τους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τώρα, κάτι ακόμα. Το τουρκικό μοντέλο φυσικά δεν μπορεί να ισχύσει στη δική μας περίπτωση. Το κόμμα μας, το Νάχτα, δεν ακολουθεί το τουρκικό πρότυπο για λόγους που είναι καθαρά συνταγματική. Η Τουρκία είναι μουσουλμανική χώρα αλλά δεν είναι αραβική χώρα. Είναι η μόνη χώρα όπου ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους βρίσκεται μέσα στο Σύνταγμα, ενώ αυτό δεν ισχύει για τι δικέ μας χώρες. Και το Ισλάμ είναι με έμεσο ή άμεσο τρόπο κρατική θρησκεία. Επομένως η Νάχτα δεν ακολουθεί το τουρκικό ε, πρότυπο. Το ξέρουν πια οι Τούρκοι συναδελφοί μας ξέρουν ότι έχει χωριστεί το μοντέλο του κράτους με, το, με, τον με την Ισλαμική θρησκεία και αν δει και τις δηλώσεις του κυρίου Εντογάν πρόσφατα για τις αμβλώσεις βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφή. Η Νάχτα χρησιμοποίησε αυτή την ε, φρασιολογία γιατί απλώς θέλανε να την εκμεταλλευτούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ομιλητών. Αφού υπενθυμίσω στους εμπειρογνώμονες μας ότι πρέπει να κρατήσουν το όριο αυτό των δεκαλευτών για τις παρεμβάσεις τους για να υπάρχει αρκετός χρόνος και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Έχουμε λοιπόν τρία άτομα στο πάνελ, το δεύτερο πάνελ, την κυρία Ναμπία Χαντούς, από τη Δημοκρατική Ένωση Γυναικών του Μαρόκου. Είναι πανεπιστημιακή κυρία Χαντούς και σύμβουλος στα θέματα ισότητας δικαιωμάτων των φύλων. Ανήκει σε διάφορες οργανώσεις που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών όπως είναι το δίκτυο Ευρωμεσογειακό για τα δικαιώματα των γυναικών και έχει μεγάλη πείρα σε συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, μετέχει στον Αραβικό Σύνδεσμο και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Δεύτερο μέλος του πάνελ είναι ο δόκτωρ Χόντα Μπαντράν, που είναι ο πρόεδρος ή πρόεδρος της ε, Ένωσης για τις ε, Γυναίκες της Αραβίας στην Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα Αιγυπτιακό φορέα ο οποίο δουλεύει σαν γενική αιγίδα φορέων και συμμετέχει σε ενέργειες με άλλους φορείς για να δώσει στις γυναίκες βασικές πτυχές ασφάλειας σε συνεργασία με διάφορους διεθνούς οργανισμούς μέσα στα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και πρωτού δώσω το λόγο στην κυρία Εστρέλα, θέλω να παρουσιάσω και την κυρία Σόφη Μπέσης, από, τον, τη Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία είναι αναπληρώτρια γενικός γραμματέας από την Τινησία, αυτού του φορέα της Διεθνούς ε, Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ερευνήτρια στο Ίδρυμα Στατηγικών Μελετών στο Παρίσι και εργάζεται σε θέματα ανάπτυξης στην, ε, στον αραβικό χώρο. Έχει δημοσίευσει πολλά βιβλία για τις γυναίκες στον αραβικό χώρο και άφα και θα ήθελα λοιπόν να δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Χάντους, την κυρία Νάμπια Χάντους. Donc, en réalité, parler Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση του Μαρόκου και θα, το, θα θέλαμε να το δούμε αυτό σε κάποιο βάθος χρόνου, μέσα σε ένα διάστημα 10-15 χρόνων. Γιατί για το Μαρόκο υπήρξαν πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ξεκίνησαν και θα χωρίσω την παρέμβασή μου σε δύο τμήματα. Υπήρξαν δύο χρονικές περίοδοι στις οποίες θα αναφερθώ. μεταρρυθμίσεων, δύο γενιές μεταρρυθμίσεων, Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με τη, μεταβατική μετα... με τη δημοκρατική μετάβαση από το 1998 που έγινε η πολιτική μετάβαση είναι μια χρονική περίοδο που γνώρισε μια θα έλεγα θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών και η οποία είχε και κάποια διάρκεια. Και τώρα πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι αυτό το οποίο συνέβαλε σε αυτή τη θετική εξέλιξη, το ότι υπήρξε μια πραγματική δημοκρατική μεταξέλιξη, μια θέληση για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών και ένα κίνημα γυναικών το οποίο πήρε επαγγελματικό χαρακτήρα που συσσόρευσε πολλή εμπειρία και είναι ένα σώμα το οποίο μπορεί να καταθέτει προτάσεις και όχι απλώς να κινητοποιεί τις γυναίκες. Και κάτι το οποίο χαρακτήρισε αυτή την περίοδο ήταν η προσέγγιση στην εργασία για τα θέματα αυτά. Η χρήση των ενώσεων, κοινωνίας των πολιτών. Και υπήρξαν και πτυχές που ευνόησαν τη συμμετοχική δημοκρατία. Ήταν συμμετοχικές πρωτοβουλίες. Υπήρξαν δηλαδή πρωτοβουλίες που πέρασαν μέσα από επιτροπές που συμμετείχαν εκεί και άνδρες και γυναίκες, συμμετείχαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Η τελευταία τέτοια διαδικασία είχε να κάνει με το Σύνταγμά μας, το οποίο εξεπονήθη με μια διαδικασία συμμετοχή, η οποία λαμβάνει υπόψη και το σφιγμό και τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών. Το κράτος δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά είναι σε επαφή και διαβουλεύεται με την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε λοιπόν μέσα σε ένα πρώτο πλαίσιο το οποίο ήταν αυτό της πολιτικής εναλλαγής το, από το 1998 και οδήγησε στην πρώτη γενιά μεταρρυθμίσεων που οδήγησε σε σημαντικές προόδους σε ό,τι αφορά το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο και επίσης σε σχέση με την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών εν γέννη, αλλά επίσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι μεταρρυθμίσει ήταν αυτέ. Ήταν κυρίω σε νομοθετικό επίπεδο. Μεταρρυθμίσεις μίζωνος επίπεδου, μεταρρύθμιση του αστικού κώδικα. Μιλάμε για οικογενειακό κώδικα πλέον και όχι για το καθεστώς του κάθε ατόμου το οποίο έβαζε τις γυναίκες σε υποδέστερη θέση. Είναι λοιπόν ένα νέο οικογενειακό κώδικα, ο οποίο δίνει δικαιώματα στι γυναίκε και τα παιδιά. Επίση, ο εργασιακό κώδικα και ο ποινικό κώδικα που μεταρρυθμίστηκαν το 2003 με κάπω συνοπτικό τρόπο, ήταν απλώ ορισμένε διατάξει που άλλαξαν. Και ο κώδικα ηθαγένεια που άλλαξε το 2007, που δίνει τη δυνατότητα στην μαροκινή γυναίκα να μεταβιβάζει, να προσδίδει την ηθαγένειά ε, τη στα παιδιά τη. Αυτές είναι λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες άλλαξαν και την οτροπία των ε, πολιτών στο, στη χώρα μας. Γιατί με την νομοθεσία αυτή αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματα των γυναικών. Το Μαρόκο επίσης έχει αναλάβει δεσμεύσεις σε εθνικό όπως και σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε μια, μια διαδικασία θεσμικής νομιμοποίησης της ισότητας των γυναικών και των ανδρών στο δημόσιο χώρο, αλλά επίσης και μια σειρά πολιτικών κατατομής. Ξεκίνησε σε τέσσερα ή πέντε υπουργεία, σε θέματα εθνικής εκπαίδευσης, επικοινωνίες κτλ. αυτές τις διαδικασίες. Και όλα αυτά έγιναν μέσα από σχέδια μαζί με εταίρους μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πρόκειται απλώς και μόνο για σχέδια, αυτό σημαίνει ότι δεν ενσωματώνονται πλήρως στην πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Επίσης έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει μια εθνική στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών και μια ατζέντα της κυβέρνησης του 2011 ώστε η ισότητα αυτή να επιτευχθεί και στην πράξη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο κύριος χρηματοδότης. Υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά τελικά έχει υποστηριχθεί αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλαβαν χώρα αλλαγές σε επίπεδο λιπτών απόφασης στα πλαίσια της κυβέρνησης. Αλλά αν είναι μια στρατηγική του κράτους του Μαρόκου και όχι απλώς μιας κυβέρνησης, θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον. είχαμε και την ε, διαδικασία πρόθεσης μιας κουλτούρας ισότητος με τα εθνικά σχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που και αυτή υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δεύτερη διαδικασία είναι η των επιφυλάξεων. Όπως ξέρετε το Μαρόκο για πάρα πολλά χρόνια από το 2008 μέχρι το 2011 ανακοίνωσε ότι ήρε τι επιφύλαξης του mm -hmm. σε σχέση με τη σύμβαση του Σεντάν και αυτό τελικά έλαβε χώρα στις 7 Απριλίου του 2011. Αυτά λοιπόν έγιναν μέσα και στην διαδικασία της Αραβικής ε, Άνοιξης. Ήταν μέσα στα πλαίσια ενός αγώνα για την ε, ε, ισότητα των γυναικών, η λεγόμενη Άνοιξη Ισότητος. Υπήρξε λοιπόν η άρση των ε, επιφυλάξεων και η προσχώρηση στο προαιρετικό πρωτόκολλο που αφορά το λαθρεμπόριο ανθρώπων και ιδίω γυναικών. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ώστε να κυρωθεί η προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση αυτή. Έτσι έκανε σημαντικά βήματα λοιπόν το Μαρόκο για την προσχώρηση σε αυτή τη συνθήκη. Τρίτον, υπήρξαν πάρα πολλά μέτρα για να ξεπεραστούν ορισμένε μορφές διακρίσεων, φυσικά όχι όλες οι διακρίσεις. Μπορώ να σας πω εδώ απλώς για τις γυναίκες που βρίσκονται στα εδάφη συλλογικής καλλιέργειας και πρόκειται για γέες που δίδονται από το αρμόδιο Υπουργείο σε άτομα ή σε ε, εταιρείες για να γίνει μια επέκταση των αστικών συνοικισμών. Έχουμε από το 1919 μια εγκύκλιο για τα θέματα αυτά που επιτρέπει απλώς και μόνο τη δυνατότητα να αποζημιώνονται οι άνδρες σε μία φυλή αλλά όχι οι γυναίκες. Εμείς στην Δημοκρατική Οργάνωση Γυναικών του Μαρόκου έχουμε εργαστεί με τις γυναίκες αυτές οι οποίες διεξεδίκησαν το δικαίωμα να αποζημιούνται και αυτές οι ίδιες. Να έχουν μια ίση λοιπόν δυνατότητα αποζημίωσης και από το 2010 αρχίζει πλέον να ισχύει η δυνατότητα αποζημίωσης των γυναικών σε ίσο επίπεδο με τους άντρες. Για πρώτη φορά λοιπόν θεωρούνται ότι έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας αυτών των γεών όπως και οι άνδρες και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Γιατί για τις αποσημειώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το κληρονομικό δίκαιο, δηλαδή μία μερίδα για τους άνδρες και μισή μερίδα για τις γυναίκες, απλώς εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία που εφαρμοζόταν διαδικασία αυτή που απέκλειε τις γυναίκες και για μας είναι πραγματικά μια σημαντική πρόοδος που μας επιτρέπει να μην αποκλείονται οι γυναίκες και να μπορούμε να διεκδικήσουμε την ισότητα. Υπάρχει βέβαια το θέμα της ερμηνείας αυτών των κειμένων. Αλλά υπάρχουν και πιο σύγχρονες ερμηνείες που αντικρούν την αρχική αντιμετώπιση στα θέματα αυτά. Επίσης, το κίνημα των γυναικών στο Μαρόκο θεωρούμε τα κεκτημένα μας δεν είναι δεδομένα, είναι εύθραυστα αυτά τα κεκτημένα. Παραδείγματο χάρη στον οικογενειακό κώδικα δεν υπήρξε συνολική μεταρρύθμιση του οικογενειακού κώδικα. Παραμένουν πάρα πολλέ διατάξει οι οποίε έχουν διακριτικό χαρακτήρα κατά των γυναικών και θα πρέπει να εργαστούμε για να τι διαγράψουμε. Παραδείγματο χάρη ο κώδικα ηθαγένεια και αυτό έχει τα ίδια στοιχεία. Δόθηκε δυνατότητα στη γυναίκα να δίνει την ηθαγένειά της στα παιδιά της όταν είναι παντρεμένη με ένα ξένο αλλά δεν μπορεί να δώσει ποτέ την ηθαγένειά της στον άντρα της. Ενώ ο άντρας μπορεί να δώσει την μαροκινή εθνικότητα και στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδου διατάξει για τι οποίε πρέπει ακόμα να ασχοληθούμε και να αγωνιστούμε. Μέχρι το 2011 επίσης Υπήρχαν ακόμα πολλέ διακρίσει, είχαν υπάρξει πρόοδοι για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά όλα αυτά δεν επαρκούν ακόμα. Από το 2011, όταν ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, το Μαρόκο πέρασε σε μια δεύτερη γενιά μεταρρυθμίσεων. Από τη στιγμή που υπήρξε ο λόγος του βασιλέως, ο οποίος ε, Διεκήρυξε την συνταγματική μεταρρύθμιση στο Μαρόκο, ενός συντάγματος το οποίο υπήρχε από το 1968 και το οποίο σύνταγμα περιείχε πολλές διατάξεις δημοκρατικού χαρακτήρα μέσα σε εισαγωγικά, ίδιο στον πολιτικό χώρο, αλλά συγχρόνως σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των γυναικών ένα προήμιο μονάχα, το προήμιο μονάχα του παλαιού συντάγματος μιλούσε για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση, του δικαιώματος στην υγεία, στη στέγαση και όλα αυτά. Δεν ήταν ιδιαίτερα σαφή όλα αυτά. Δεν υπήρξε αναφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τα κατανοούμε σε διεθνές επίπεδο. Δεν υπήρχε απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν υπήρχαν άθρα που να αφορούν άμεσα την ισότητα και την καταπολέμηση της ανισότητας. Μετά όμως από το λόγο του βασιλέως άρχισαν οι προσπάθειες τροποποίησης του συντάγματος. Οι οργανώσεις των γυναικών όπως και όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ξεκίνησαν τις ενέργειές τους για να υπάρξει ένα νέο συντάγμα, ένα σχέδιο νέου συντάγματος το οποίο συζητήθηκε και σε μια επιτροπή η οποία έχει ευρύ εκπροσώπηση με άνδρες, γυναίκες, εκπροσώπους ε, ανθρωπινών, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεων γυναικών, οργανώσεων αγωνιζομένων για τα πολιτιστικά δικαιώματα, όπως ήταν η που είναι τα Υπήρχαν αρμόδιοι για τα συνταγματικά θέματα και τα λοιπά. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα μνημόνιο Υποβλήθηκαν και άλλα υπομνήματα αυτού του είδους από οργανώσεις γυναικών, ιδίως για τα δικαιώματα των γυναικών. Ο στόχος μας λοιπόν να μην αντιμετωπίσουμε το σύνολο του συντάγματος. Το υπόμνημά μας λοιπόν, το μνημόνιμο όμως, το οποίο μπορώ να σας δείξω αν θέλετε, αντιμετώπισε το, το γενικό πλαίσιο και τις ιδιαίτερες διατάξεις και υπήρξαν πολλές προτάσεις οι οποίες πέρασαν στη συνέχεια, έγιναν δεκτές όπως είχαμε διατυπώσει, γιατί είχαν τη σωστή διατύπωση. Και επομένω εξασφαλίστηκε με τον τρόπο αυτό ότι πολλές από τις διατάξεις του υπομνήματός μας έγιναν δεκτές είτε στο προήμιο του συντάγματος είτε μέσα στα άρθρα και το νέο σύνταγμα στο άρθρο 19 αναφέρεται στην ισότητα και στην μη εφαρμογή διακράσεων με την εφαρμογή επίσης και μιας αρχής η οποία εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων. Η συνταγματική λοιπόν μεταρρύθμιση έλαβε χώρα, γίναμε ακουστές από την Επιτροπή αυτή για τα θέματα αυτά συνταγματικά, αυτό ήταν πολύ θετικό. Θεωρήσαμε ότι αυτό το νέο σύνταγμα είναι ένα σύνταγμα για όλους και όλες. Δεν είναι ένα σύνταγμα απλώς το οποίο υποστηρίζει ένα κράτος, μια κυβέρνηση. Ήταν ένα σύνταγμα το οποίο μπορούσε να αντανακλά τις επιδιώξεις, τις προσδοκίες όλων των Μαροκινών. Αναγνώριζε τουλάχιστον την υπεροχή των διεθνών συμβάσεων επί του Μαροκινού δικαίου, αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, καταγράφει μια σειρά από αρχές σε σχέση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλα αυτά οδηγούν προς μια ουσιαστική θέση του πολίτη, γιατί όπως είπε και η συνάδελφός μας από την Τινησία, δεν έχουν ουσιαστική ηθαγένεια οι γυναίκες στο Μαρόκο, γιατί υπάρχουν πολλές νομοθετικές διατάξεις που είναι διακριτικού χαρακτήρα και πολλά δικαιώματα στα οποία δεν έχουν πρόσβαση ακόμα. Λοιπόν, καθιερώνεται η ισότητα εδώ και γυναικών στο δίκαιο, το αστικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, το πολιτιστικό, αναφέρεται η έννοια της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Αναγνωρίζεται και η θετική δράση. Για πρώτη φορά δεν πρόκειται να μας πούν ότι μία ποσόστοση παραδείγματος χάρη στις εθνικές λίστες για τις βουλευτικές εκλογές δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνταγματικό. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε να υπάρχουν ποσοστώσεις για τις γυναίκες. Μέχρι τώρα το Μαρόκο είχε μονάχα εθνικά ψηφοδέλτια τα οποία περιλάμβαναν ένα αριθμό εδρών που ήταν για τις γυναίκες αλλά αυτό ήταν με την θέληση των πολιτικών κομμάτων και μόνο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα που να υποχρεώνει ένα πολιτικό κόμμα να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Το κάναν μονάχα από την δική τους πρωτοβουλία. Ο νέος θεσμικός μηχανισμός λοιπόν για το σεβασμό και την προ... προώθηση των δικαιωμάτων περιλαμβάνει και ένα διαμεσολαβητή ο οποίος ε, θα αναλάβει μάλλον την ευθύνη για την ισότητα. Υπάρχει μια άλλη αρχή για την ισότητα και τον αγώνα κατά κάθε μορφής διακρίσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του νέου συντάγματος και το άρθρο 164 του συντάγματος και υπάρχει και ένα συμβουλευτικό συμβούλιο για την οικογένεια και την παιδική ηλικία. Εκεί υπάρχει μια διαφορετική ίσως απόχρωση από και το πώς το βλέπουν αυτό οι Ισλαμιστές που το βλέπουν στα πλαίσια της ε, μουσουλμανικής οικογένειας. Υπάρχουν διαφορές απόψεις να υπάρχει περιπτώσει ένα συμβουλευτικό συμβούλιο ανεξάρτητο το οποίο καλύπτει όλο το Μαρόκο. Δεν μπορούμε... να πούμε βέβαια ότι έληξε ο αγώνας αυτός η προσπάθεια, αλλά έγιναν σημαντικές πρεότητες. Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, ε, δεν έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις στο κείμενο. Υπάρχει και η νομολογία, το Σύνταγμα δεν μας λέει πού πρέπει ακριβώς να βασιστούμε και η νομολογία είναι βασικά μια νομοθεσία που προέρχεται βασικά από τη Σαρία αλλά και από τις διεθνείς συμβάσεις. Υπάρχει εδώ, υπάρχουν δύο πηγές. Η εφαρμογή των ρητρών είναι προβληματική διότι καμιά φορά δεν γίνεται με σύγχρονο τρόπο δηλαδή. Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο για, την, για τα οικογενειακά θέματα έχει προβλήματα. Α, δεν έχουμε χρόνο. Καλά, λοιπόν. Έχουμε ακόμη πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Είναι η τελευταία διαφάνεια εδώ. Δηλαδή, ο αγώνας μας για την ισότητα ανδρών και γυναικών συνεχίζεται και με κάθε ευκαιρία κινητοποιούμαστε και κινητοποιούμε για να διατυπώσουμε αιτήματα ή να κάνουμε συστάσεις. Ζητήσαμε από τον καινούργιο Πρωθυπουργό να πάρει μέτρα, από τον Υπουργό Οικογενειακών Θεμάτων κλπ. Δηλαδή δεν σταματάμε πουθενά. Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο Μαρόκο δεν έχουν ακόμα καταλήξει να λύσουν το θέμα των ίσων δικαιωμάτων. Θα σας πω τι μένει ακόμη να γίνει. Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες για Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό μπορεί να γίνει ήδη. Γιατί το κράτος το έχει προβλέψει. Η εφαρμογή του προγράμματος ισότητας είναι άλλος αγώνας όμως σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εδώ ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε. Και η εφαρμογή του θεσμικού προγράμματος για την ισότητα είναι το τρίτο θέμα για να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή της, στρατηγικής, της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα. Το Εθνικό Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς το παρόν συζητάει το άρθρο 19 του Συντάγματος για την άρνηση, καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης στην αρχή συζητούσε αν η διακριτική μεταχείριση αφορά κυρίως ή μόνο τα φύλλα, αλλά τελικά δεν είναι τελείωσε η συζήτηση αυτή. Δεν νομίζω ότι μακρηγόρησα ή κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αν υπάρχουν άλλες απορίες, ευχαριστούμε πολύ κυρία Χαντούς για τις πληροφορίες σας αυτές για την κατάσταση των γυναικών στο Μαρόκο αν δεν απατώμε. Θα συνεχίσω στα Πορτουγαλικά δίνοντας το λόγο στην κυρία Όντα Μπαντράν. Ορίστε κυρία μου. E και να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να κάνω κάποιες συστάσεις να ζητήσω στους ε, ειδικέ μας να περιοριστούν στα 10 λεπτά. 10 λεπτά που έχουν προβληθεί για την παρουσίαση των εισηγήσεών τους, γιατί έχουμε καθυστερήσει αρκετά και Επίσης να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έγιναν και που θα γίνουν υπάρχουν και στο ίντερνετ. Έχουμε κάποιους που έχουν ζητήσει το λόγο για να παρέμβω. Θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ όσο γίνεται καλύτερα, ε, ώστε να εκπροσωπηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πρώτα ζήτησε το λόγο η κυρία Κάρμεν Ρομέρο Λόπες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ το κοινοβούλιο αυτό... Εργαζόμαστε σε διάφορες ε, επιτροπές ταυτόχρονα και εμείς που είμαστε εδώ παρούσες έχουμε και δουλειά ταυτόχρονα αλλού. Εγώ στις 5.30 πρέπει να είμαι αλλού ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων γιατί θα είναι εκεί ο Μπεντζαφάρ και θα μιλήσει για τη κατάσταση ε, προόδου στη συνταγματική συνέλευση της Τινησίας. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ρόλος των γυναικών, ποιος θα είναι ο μελλοντικός εκλογικός ε, νόμος, ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν, τα οποία μας επηρεάζουν ως γυναίκες και ως ευρωβουλευτές. Είναι κρίμα που πρέπει να είμαι εκεί λοιπόν στις 5.30, γι' αυτό και ζήτησα το λόγο τώρα να δω αν μπορούσαμε να διακόψουμε λίγο το δεύτερο αυτό πάνελ, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσω να πάρω το λόγο. Ναι, μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Εγώ θέλω να είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε, γιατί πραγματικά μετά από τις δύο πρώτες παρεμβάσεις που ήταν τόσο διαφορετικές, τελικά κατέληξα ότι σε αυτές τις χώρες ε, η κατάσταση είναι και τελείως διαφορετική. Και εμείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να γνωρίζουμε πιο συγκεκριμένα κάθε μία από αυτές τις χώρες. Το να μιλάμε γενικά για Βόρεια Αφρική σημαίνει άγνοια. Γιατί πραγματικά κάθε χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της και θα έπρεπε να γνωρίζουμε πιο βαθιά την κατάσταση της κάθε χώρας. Επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής για το Μαγκρέπ, πιστεύω πως τώρα η Επιτροπή μας θα έπρεπε να διοργανώσει αυτές τις ακροάσεις πάντα σε συνδυασμό με την αντιπροσωπεία του Μαγκρέμπ ή με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Γιατί πραγματικά θα ήταν πιο αποτελεσματική η δουλειά μα. γιατί θα συντονίζαμε καλύτερα τη δουλειά μα. Είναι θέμα συντονισμού. κυρία συνάδελφος που ήταν στην επιστολή παρατήρησης των εκλογών πήγε εκεί, ναι, έκανε έκθεση σχετικά με στην Επιτροπή Εξωτερικών, στην, Επιτροπή, στην, στην Αντιπροσωπεία για το Μαγκρέμπ. Υπάρχουμε πολλοί που δουλεύουμε για αυτά τα θέματα, αλλά όμως καθένα χώρια. Ενώ θα έπρεπε να γίνονται πιο συντονισμένε κινήσεις, ώστε να είναι και πιο αποδοτική η δουλειά μας. Η παρέμβασή μου λοιπόν ήταν βασικά για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε καλύτερα την κατάσταση σε κάθε μια από τις χώρες και στη συνέχεια για να μπορούμε να κάνουμε μια ανακρόαση με μια ευρύτερη επιτροπή και όχι μόνο με την αντιπροσωπεία του Μαγκρέβ αλλά και με την, αντιπροσωπή, την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όπου θα έπρεπε να αναμειχθεί γιατί δεν είναι μόνο υπόθεση των γυναικών αυτή αλλά είναι υπόθεση όλων των Ευρωπαίων και όλων των ε, χωρών της Μεσογείου και των πολιτών τους. Να κλείσω λέγοντας μόνο γιατί πραγματικά με συγκίνησε το θέμα της Λιβύης. Φυσικό είναι να συγκινείται κανείς γιατί το θέμα της βίας, της βίας κατά τη διάρκεια πολέμου, αλλά η βία είναι κάτι το οποίο είναι οριζόντιο ε, επηρεάζει όλες τις γυναίκες. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, να στηρίξουμε τις γυναίκες της Λιβύης για να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Και οι τινήσιες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, ώστε να αναγνωριστούν ως θύματα ε, του πολέμου. Είναι απαραίτητο. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει πιο εις βάθος δουλειά εδώ και να δουλέψουμε ως ευρωβουλευτές και για το, Ευρωπαϊκό δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να δώσουμε την πολιτική μας στήριξη σε κάθε μία από όλες τις γυναίκες αυτές, έχοντας μια διαρκή επαφή και καλύτερη γνώση για την κατάσταση. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όπως σας είπα πρέπει να είμαι στο στο. Ε, παρουσία του Μπεν Τζαφάρα στην άλλη επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε τις διάφορες υποχρεώσεις που έχουμε, τις ε, πολυάριθμες ταυτόχρονες συνεδριάσεις. Δεν είναι εύκολο σίγουρα. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλα αυτά τα θέματα τόσο σε τούτη την Επιτροπή όσο και στις άλλες γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και πολύ επίκαιρο. Όλοι μας ε, παρακολουθήσαμε με μεγάλες προσδοκίες την ε, Αραβική Άνοιξη και δώσαμε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο που παίζουν οι γυναίκες και που συνεχίζουν να οικοδομούν τη δημοκρατία στις διάφορες χώρες. Είναι προς το συμφέρον μας να συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα αυτό και να ε, παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Χόντα Μπαδράν. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την Επιτροπή που κάνει αυτή την ακρόαση και που με κάλεσε. Ίσως να είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσω αυτό το μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα για την εξαίρετη εισαγωγή που κάνατε για τις χώρες μας. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή λίγο του χρόνου σε κάποια θέματα. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο πρόσφατα δημοσίευσα στη... Εδώ σας το δείχνω. Αν κανείς θέλει να εμβαθύνει, πρόκειται για την τελευταία εκδοσή αυτού του περιοδικού. Εγώ επέλεξα αυτό τον τίτλο διότι Ανακαλύψαμε στη χώρα μας ότι το θέμα είναι αγώνας εξουσία στην ουσία ε, και η οργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντικό συστατικό σε, αυτές, σε αυτόν τον αγώνα για την εξουσία, ώστε να μπορούμε να είμαστε δυνατές. Κοιτάξτε πόσος κόσμος τώρα σε αυτή τη δεύτερη διαφάνεια στην πλατεία Ταχρήρ. Πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος ήρθε στην πλατεία. Μάλιστα η Ταχρήρ θα, θα πει απελευθέρωση. Έχει νόημα ε, το όνομα της πλατείας και γι' αυτό και οι νέοι θέλαν να συναντηθούν στην ε, πλατεία ελευθερίας στην ουσία γιατί σήμαινε ότι θέλαμε να ελευθερώσουμε τη χώρα μας από το ε, ε, δικτατορικό καθεστώς. Πολλοί κόσμος, πολλές γυναίκες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταχρήρ λοιπόν στην Πλατεία Ελευθερίας αλλά και σε άλλες πλατείες ολόκληρη τη χώρα οι γυναίκες στην ουσία ζητούσαν τα ίδια πράγματα όπως οι άνδρες και οι κοινέοι ζητούσαν ισότητα, ζητούσαν δικαιοσύνη, ζητούσαν δημοκρατία. Δεν υπήρχαν ε, χώρια αιτήματα για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Και υπήρχαν ένα, ε, γυναίκες από όλες τις ε, τάξεις, γυναίκες ε, πιο ηλικιωμένες, ορισμένες με φερετζέ, χωρίς, όλα. Και εκεί όχι μόνο κρατούσαν πάνω, αλλά έκαναν και παραπάνω πράγματα ακόμα. Ε, φρόντιζαν τους αρρώστους και τους τραυματίες, μοίραζαν φαγητό, καθάριζαν το πρωί μετά ε, αφού είχε συγκεντρωθεί είχαν συγκεντρωθεί βρωμιές στην πλατεία. Εμείς λοιπόν συμμετείχαμε ως άτομα, εγώ, το επιτελείο μου, η οικογένειά μου, ήμασταν όλοι εκεί, αλλά συμμετείχαμε και ως μικιο μοιράζαμε κουβέρτες γιατί ήταν χειμώνα και έκανε κρύο και έπρεπε να περάσουμε όλη τη νύχτα στις πλατείες. Ε, επίσης ε, μοιράζαμε φάρμακα. Συμμετείχαμε λοιπόν ως άτομα, α, ως ε, φεμινιστικές ε, και ως φεμινιστικές ΜΚΟ στην Επανάσταση. Έπειτα περάσαμε στη μετάβαση στην δημοκρατία και έφνης, αφού ενώ ήμασταν ε, πραγματικά εταίροι μας ε, διώξαν, μας απόκλεισαν από οποιονδήποτε μηχανισμό, από οποιαδήποτε επιτροπή, από οποιοδήποτε γεγονός, εκδήλωση. Για παράδειγμα, φτιάχτηκε μια επιτροπή για να διατύπωση κάποιον από τα άρθρα του συντάγματος, ούτε μια γυναίκα δεν ήταν σε αυτήν την επιτροπή. Όχι γιατί δεν υπήρχαν γυναίκες, γιατί έχουμε μια γυναίκα που είναι αντιπρόεδρος του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Μπορεί κανείς να διερωτηθεί γιατί αυτή η γυναίκα δεν προσεκλήθη, γιατί το Στρατιωτικό Συμβούλιο, το ανώτατο Συνταγματικό Συμβούλιο ανέλαβε την εξουσία και όλοι ξέρουμε ότι τι, τι, τι θα πει αυτό. Δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τις γυναίκες ως ίσους ισότιμους εταίρους να κάθονται στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων, συζητήσεων κτλ. Είναι τελείως πατριαρχικό σύστημα, τελείως αρσενικό σύστημα. Ο φεμινισμό είναι κατά του στρατού, γιατί αν θέλει κανεί να είναι αξιωματικό ή στρατιώτη, θα πρέπει να είναι σκληρό, να είναι ε, αρενοπό, να μην είναι θηλυκό, θηλυπρεπή, να μην είναι αδύναμος και ούτω καθεξής. Και δεν ήταν μόνο το στρατιωτικό συμβούλιο το οποίο ορθώθηκε εναντίον μας, αλλά ξαφνικά ολόκληρη η πολιτική, όλα τα πολιτικά ισλαμικά ε, κόμματα, ομάδες επέστρεψαν από τη Σαουδική Αραβία, από τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, όπου ερμηνεύεται το Ισλάμ με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Η πιο αυστηρή ερμηνεία κατά των γυναικών δίνεται στις χώρες αυτές. Πριν ακριβώς από την, την ε, Επανάσταση υπήρχε ένας ανταγωνισμός κατά των γυναικών, διότι υπήρχε μια σύνδεση ανάμεσα στα λίγα πράγματα που είχαν επιτύχει οι Αιγύπτες γυναίκες και τη Σουζάνα Μουμπάρακ που ήταν η σύζυγος του Προέδρου και η οποία θεωρεί το τμήμα της διαφθοράς και όλων. Ακόμα αρχίσανε να την κατηγορούν αυτήν λες και όλα εξαιτία της γίνανε. Λες και όλα αυτή τα έκανε η Σουζάν Μουμπάρα και όχι ο σύζυγός της ή ολόκληρο το σύστημα που ήταν διεφθαρμένο. Λόγω όλων αυτών όπως σας είπα αποκλειστήκαμε. Μας βάλανε στην άκρη. Και όχι μόνο αυτό. Ασκήθηκε βία και χειδεότητα. Μπορείτε να δείτε αυτή την περίφημη εικόνα του κοριτσιού με το θαλασσί σουτιέν. Οι στρατιώτες πραγματικά την έριξαν κάτω. Και, ότι, και είπαν ότι μόνη της γδύθηκε, ε, αλλά δεν το κάναμε εμείς. Και σίγουρα θα ακούσατε και για τα τεστ ε, παρθενίας. Το Στρατιωτικό Συμβούλιο απλά και μόνο για να ταπεινώσει κάθε γυναίκα που βγήκε στους δρόμους και στις πλατείες της ε, υπέβαλε, υπέβαλε γύρω στα 20 κορίτσια σε τεστ παρθενίας για να δουν αν είναι ακόμα παρθένες ή όχι. Και αυτοί που τα κάναν αυτά, μετά ένα από τα κορίτσια μάλιστα τόσο πολύ γενναία ήταν που τους ε, ε, κατήγγειλε, το στρατικό συμβούλιο, αλλά τελικά όλοι όσοι ήταν του στρατού αθώθηκαν. Μετά γίνανε οι βουλευτικές εκλογές που κυριαρχήθηκαν από τα Ισλαμικά κόμματα και ομάδες. Γιατί τα υπόλοιπα φιλελεύθερα κόμματα ήταν αδύναμα. Μόνο 2% των γυναικών ε, λοιπόν έγιναν βουλευτές. Και γιατί ξαφνικά το σύστημα ποσόστοσης ε, που ίσχυε πριν από την Επανάσταση για τις γυναίκες καταργήθηκε. Ναι. Μια άλλη εκλογική νομοθεσία εκδόθηκε και ίσχυσε που ζητούσε κάθε πολιτικό κόμμα να βάλει τουλάχιστον ένα, μια γυναίκα στα ψηφοδελτιά της. Και βέβαια οι γυναίκες ήταν στο κάτω-κάτω μέρος των ψηφοδελτίων, οπότε δεν εξελέγησαν. Περίπου 75% λοιπόν των εδρών αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο μας καλύπτονται από την αδελφότητα των τους αδελφούς μουσουλμάνους και τους σαλαφιστές. Δεν ξέρω πώς μας προέκυψαν οι σαλαφιστές, εμείς δεν τους είχαμε ακουστά, αλλά ξαφνικά αν πας ε, ε, στο Αιγυπτιακό αεροδρόμιο, στο, στο, στο αεροδρόμιο θα δεις εκατοντάδες να έρχονται από τον Περσικό και από αλλού. Αυτό έτσι έγιναν τα πράγματα. Θετικά τώρα στοιχεία. Οι φεμινιστικές ομάδες και ΜΚΟ πραγματικά ξυπνήσαμε, ανησυχήσαμε και είδαμε ότι είμαστε πολύ αδύναμες ε, στην κοινωνία όσον αφορά αυτή την, τον αγώνα για την εξουσία. Γιατί στην ουσία είναι ένας αγώνας, μια μάχη. Και Είπαμε, εντάξει λοιπόν, τι, πόρους, ε, τι, τι, πηγές εξουσίας έχουμε. Θεωρητικώς η εξουσία προέρχεται από τρεις ε, πηγές. Από την ο μέγεθος της ομάδας, ε, από την καλή οργάνωση και από τους πόρους. Ευτυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτό και αν οργανωθούμε και αποφασίσαμε ότι έπρεπε να οργανωθούμε. Ο πρώτο συνασπισμός γυναικών δημιουργήθηκε, ήμασταν 16-17 φεμινιστικές ΜΚΟ, Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν και αρχίσαμε να υποβάλλουμε τίματα, να κάνουμε, αρχίζουμε διαδηλώσεις στους δρόμους και στις πλατείες και κάναμε διαμαρτυρίες λόγω των ε, τεστ παρθενίας και της ε, απόφασης τιμιγορίας αθώ, αθώωσης των ε, υπευθύνων. Ακούσαμε πολλές επικρίσεις ότι το κίνημα το γυναικείο είναι λιτίστικο. Εμείς αποφασίσαμε λοιπόν ότι δεν θα είμαστε πια μια ελίτ, θα μπούμε, θα κατέβουμε στο, μέχρι το τοπικό επίπεδο. Και αυτό και κάναμε και για πρώτη φορά οργανώσαμε διάσκεψη που παρακολουθήθηκε από 3.000 εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Δεν ήταν μόνο τα φεμινιστικά κινήματα, γιατί δεν θέλαμε να χωριστούμε από την υπόλοιπη κοινωνία των πολιτών και, και εδώ μπορείτε να δείτε, αυτό ήταν το πρώτο μας συνέδριο. Και αυτό σήμανε δύο σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, φτιάξαμε ένα χάρτη που δήλωνε ποια είναι τα αιτήματά μας και ότι πρέπει να είμαστε εταίροι και μετά την Επανάσταση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής. Και το άλλο το οποίο προέκυψε επίσης ήταν ότι έπρεπε να φτιάξουμε μια Αιγυπτιακή Φεμινιστική Ένωση. Από το 50 δεν είχαμε καμιά ε, τέτοια, τέτοιο κίνημα. Ο ήταν, είχε φτιάξει ε, ένα τέτοιο κίνημα το 32, αλλά έκτοτε, ε, μάλλον το σταμάτησαν το 50 αλλά έκτοτε τίποτα άλλο δεν είχε διοργανωθεί. Και έτσι ξεκινήσαμε ώστε να είμαστε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί και για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών ζητήσαμε από τους υποψηφίους να έρθουν να μας μιλήσουν και να μας πούνε τι έχουν σκεφτεί για τις γυναίκες. Και επειδή αρχίσαμε να έχουμε μεγαλύτερη ισχύ, ήρθαν και για πρώτη φορά αρχίσαν να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες. Αυτό είναι το έμβλημα της Αιγυπτιακής ε, Φεμινιστικής Ένωσης και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για δύο πράγματα. Πρώτον, η Ένωση φτιάχτηκε και θεσπίστηκε από κάτω προς τα πάνω. Όλοι οι, οι κυβερνήτες της Αιγύπτου συμμετείχαν στη δημιουργία αυτής της Ένωσης. Έχουμε τώρα 100 μικιό μέλη. Έχουμε ένα ε, διοικητικό συμβούλιο 15 μελές έχουμε πρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμεία. Και είναι μεγάλη μου τιμή που εγώ είμαι πρόεδρος αυτής της φεμινιστικής, αυτού του φεμινιστικής ένωσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επίγοντα πράγματα να κάνουμε. Το ένα είναι το νέο σύνταγμα, όπου απαιτούμε να είμαστε σε αυτή την επιτροπή της τεκτική και μάλιστα πολυάριθμη πολυάριθμες, τουλάχιστον 30% ζητάμε, διαπραγματεύονται μαζί μας και δηλώνουν ότι θα μας δώσουν μόνο το 10%. Εμείς λέμε όχι, εμείς δεν πάμε κάτω από το 30%. Επίσης, ε, συντάσσουμε σχέδια για κάποια άρθρα που θα πρέπει αποκλειστικά να αφορούν τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους. Έχουμε πάρει από όλα τα διεθνή, τις διεθνείς συμβάσεις, όχι μόνο το ΣΥΝΤΑΟ, αλλά και άλλες συμβάσεις που συμπεριλαμβάνουν δικαιώματα για όλους και για τις γυναίκες και από άλλες αραβικές χώρες που τα συντάγματά τους είναι καλύτερα από το δικό μας. Μάλιστα κάνουμε τώρα μια μελέτη για να φτιάξουμε μια, ένα πρόγραμμα διετές. Οι προτεραιότητες μας είναι να αλλάξουμε την, ε, το οικογενειακό δίκαιο γιατί οι διακρίσεις ε, είναι νόμιμες ε, σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο τώρα. Και έπειτα Χρειαζόμαστε ένα εθνικό πλάνο για την εκρίζωση της, ε, του αναλφαβητισμού, γιατί το ίμιση των ε, γυναικών στην Αίγυπτο είναι αναλφάβητες. Και όταν είσαι αναλφάβητος, οι αδελφοί μουσουλμάνοι ε, σε χειρίζονται, σου δίνουν μετά και εξουσιοδοτήσεις στις εκλογές και πάει λέγοντας αυτά. Αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Και τι χρειάζεται τώρα εμείς από τη διεθνή κοινότητα, να σας πω. Εμείς χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, χρειαζόμαστε και συναισθηματική στήριξη. Και τι θα πει συναισθηματική στήριξη. Οποιαδήποτε φορά κάποιοι από εσά έρχονται στην Αίγυπτο, παρακαλούμε να βάζετε τα θέματα των γυναικών στην ατζέντα όταν μιλάτε με τους υπεύθυνου ε, για την λήψη των αποφάσεων. Και να σας πω θα σας πούνε καταρχήν ότι ναι, τα έχουν όλα οι γυναίκες εδώ και ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι τα ίδια με τα δικά μας. Δεν είναι αλήθεια. Σας παρακαλώ μην το λέτε, μην τους πιστεύετε. Και όταν ε, το αναφέρονται, το αναφέρουν αυτό, θα πρέπει εσείς να το διαψεύδετε. Χρειαζόμαστε και τεχνική βοήθεια. Δεν είμαστε τέλειοι. Μαθαίνουμε από τις άλλες χώρες, ανταλλάσσοντας εμπειρίες. Χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη σας, τη δική σας που είστε μέλη σε ευρωπαϊκές ε, ΜΚΟ. Σας ε, παρακαλούμε να έρθετε και να μας δώσετε την τεχνική σας βοήθεια και τέλος οικονομική βοήθεια, διότι επίσης χρειαζόμαστε πόρους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Αιγυπτιακή κυβέρνηση σταματάει οποιαδήποτε διεθνή συνεργασία για τις ΜΚΟ και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούν να αλλάξουν κιόλα την νομοθεσία περί ΜΚΟ, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα για μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν την στήριξή σας και τελικά θέλω να σας πω μην νομίζετε, μην, μην πιστεύετε ότι πρόκειται για ξένη παρέμβαση. Θα σας πούνε κάποιοι ότι παρεμβαίνετε στα εσωτερικά της χώρας. Εγώ ήμουν, όταν ήμουν πρόεδρος για τα δικαιώματα του παιδιού, θα σας πω ότι είχαμε το ρητό ότι αν ε, τα δικαιώματα ενός παιδιού παραβιάζονται σε μια συγκεκριμένη χώρα, δεν είναι θέμα υπόθεση αυτής της χώρας, αλλά υπόθεση ολόκληρου του κόσμου. Να σας πω λοιπόν και αναλογικά ότι αν παραβιάζεται τα δικαιώματα μιας γυναίκας σε οποιαδήποτε χώρα, είναι θέμα όλων μας, όχι μόνο της Αιγύπτου, Βεβαίως σε διάφορους βαθμούς είμαστε βασικά υπεύθυνοι, αλλά όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Μπαντράν. Θα ήθελα να κάνω μερικά σύντομα σχόλια Φυσικά είναι δική μας ε, υπευθυνότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουμε υποστήριξη στις γυναίκες από την Αραβική Άνοιξη, από τις, στις γυναίκες της Αιγύπτου και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει τεχνική αρρωγή και χρηματική αρρωγή πέραν της ε, συγκινησιακής συναισθηματική υποστήριξης που δίνουμε. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική κατάσταση στην ε, Αίγυπτο. Είναι φανερό ότι δεν φτάνει να αλλάξει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών. Δεν τολμώ να πω ότι η κατάσταση της, γυναίκες, γυναίκας στην Αίγυπτο είναι χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν, αλλά τολμώ να πω ότι δεν είναι καλύτερη. Οι γυναίκες στην Αίγυπτο ήταν πάρα πολύ ενεργές, ήταν στο δρόμο, αγωνίστηκαν, δεν ήταν απλώς θεατές της ε, επανάστασης, ήταν πραγματικά ήταν φορείς της αλλαγής αλλά γνωρίζουμε και από την Ευρώπη, από τον αγώνα των γυναικών εδώ και πολλά χρόνια, ότι οι γυναίκες κυρίως είναι για να εργάζονται και όχι για να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτή είναι μια ιδέα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Οι γυναίκες είναι για να δουλέψουν, ξέρουν να δουλέψουν, αλλά συγχρόνως πρέπει να είναι και αυτές που λαμβάνουν αποφάσεις στο πολιτικό και οικονομικό στίβο και είναι εξίσου ικανές με τους άνδρες. Γι' αυτό δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να αποδεχτούμε οι γυναίκες να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Και ακόμα χειρότερα δεν μπορούμε να δεχτούμε ως Ευρωπαίοι οι γυναίκες να την χάνουν περιφρόνησης και ταπείνωσης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκε. Τούτου λεχθέντος θέλω να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπέση. η οποία θα μας μιλήσει για την κατάσταση των γυναικών στην Τινησία. Έχετε το λόγο. Αν θέλετε. merci Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα κάνω μία παρουσίαση συνοπτική, γιατί αν θέλω να τα πω εκτενώς, θα μιλάω για πάρα πολύ χρόνο, αν θέλω να παρουσιάσω το σύνολο της κατάστασης των γυναικών στο Μάγρεπ, στη Βόρεια Αφρική. Θα ήθελα να ξεκινήσω επειδή βλέπω να μειώνονται οι παρούσες, θα ξεκινήσω από το τέλος. Αυτά που θα έλεγα στο τέλος. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθαν να ακούσουν εμάς τις γυναίκες της Βόρειας Αφρικής για να έχουν κάποια επίγνωση των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν και άνδρες στους οποίους χαιρετίζω σε αυτή την αίθουσα αλλά η μεγάλη γυναικεία παρουσία στην ε, αίθουσα αυτή δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να βοηθήσει τι γυναίκε. οι άντρε πηγαίνουν εκεί που παίζονται τα σοβαρά παιχνίδια και άμα δεν είναι εδώ παρόντε, σημαίνει ότι το θέμα των γυναικών δεν λαμβάνεται ακόμα σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί, γιατί η πλειοψηφία των ανδρών δεν έχει καταλάβει ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ σε αυτή την περιοχή του κόσμου μέσα στον ανεμοστρόβιλο της Επανάστασης, το θέμα των γυναικών είναι κομβικό για τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα θέματα της δημοκρατίας χωρίς να μιλάμε για την κατάσταση των γυναικών. Πρώτον, μπορούμε να θέσουμε πολύ απλό φαινομενικά, αλλά δεν τίθεται αρκετά. Μπορεί να υπάρχει η έννοια του πολίτη της ηθαγένειας Μπορεί να υπάρχει δημοκρατία αν δεν είναι όλοι οι πολίτες ίσοι ενώπιον του νόμου. Αυτό φαίνεται θεμελιώδες, αυτό φαίνεται βασικό. Δεύτερο ερώτημα. Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια δημοκρατία, μια πραγματική δημοκρατία στον πολιτικό χώρο, αν σε όλους τους άλλους τους χώρους, στον κοινωνικό χώρο και στον χώρο της οικογένειας, εξακολουθεί να υπάρχει και να παραμένει μια βασική ανισότητα. Κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα. Στις χώρες λοιπόν αυτές που γίνεται η προσπάθεια δημοκρατίας της πολιτικής δημοκρατίας κλείνουν τα μάτια τους για τον οικογενειακό χώρο και τον κοινωνικό χώρο που υπάρχει μια κατάφορη ανισότητα. Σήμερα λοιπόν το θέμα των γυναικών στις χώρες αυτές οι οποίες είχαν ζήσει κάτω από δικτατορία για πάρα πολύ χρόνο, αλλά τουλάχιστον σήμερα για ορισμένε από αυτέ υπάρχει δυνατότητα ανοιχτού διαλόγου. Το θέμα των γυναικών είναι το επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών οραμάτων που αντιπαρατίθενται στο τμήμα αυτού του κόσμου. Το θέμα της ισότητας και το τόνισαν οι φίλες μου με ένα διαφορετικό τρόπο το θέμα της ισότητας θέτει το ερώτημα ανάγλυφα της θέσης της θρησκείας στην κοινωνία. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Εσύ νομίζω αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, λέει, θέτε στην κυρία Χαντούς. Το πλαίσιο αναφοράς είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες. Ωραία. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις γυναίκες, γιατί μιλάμε, μιλάμε για τη δημοκρατία, μιλάμε για την κοσμικοποίηση του κράτου, ε, καλύτερα του κράτους, μιλάμε για την ισότητα. Νομίζω ότι μιλάμε για θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Και εν συντομία, είναι γεγονός ότι υπήρξαν παραστατικές διαδικασίες, αλλαγές καθεστώτων σε ορισμένε χώρες, ίσως όχι σε άλλες, αλλά σήμερα, εν πάση περιπτώσει, ο αραβικός κόσμος είναι εν κινήσει. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο τώρα αυτή η κίνηση θα συνεχίσει. μετά από την επαναστατική αυτή κίνηση που έγινε, είδαμε να έρχονται στο προσκήνιο κόμματα Ισλαμικών αποχρώσεων σε χώρες όπως η Τινσία και η Ήπτος που ήταν θεαματική η πτώση της δικτατορίας όπως είδαμε για τις εκλογές στην συντακτική συνέλευση της Τινσίας υπήρξε μια σχετική πλειοψηφία γύρω στο 40% στο Ναχμπα, Ναχτα ενώ στην ε, Αίγυπτο το κόμμα το οποίο προέρχεται από τους αλαφιστές και την, τους αδελφούς μουσουλμάνους έχει περίπου τα 3 τέταρτα των εδρών. Δεν έχουμε λοιπόν ακόμα συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό το θέμα των γυναικών βρίσκεται στην, στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Τον Οκτώβριο του 2011 με την πτώση του Καντάφη, ο πρώτος επίσημος λόγος του μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου σε μια χώρα η οποία είχε εξανδραποδιστεί από 40 χρόνια δικτατορίας από εμφύλιο 9 μηνών από του βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ η πρώτη προτεραιότητα που αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του Μεταβατικού Συμβουλίου ήταν να πει ότι θα επανέλθει η Σαρία σε πλήρες επίπεδο και θα επανέλθει και η πολυγαμία πλήρως. Αυτή ήταν η πρώτη λοιπόν ανακοίνωση του Μεταβατικού Συμβουλίου. Λες και δεν υπήρχε άλλη προτεραιότητα. Λες και δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα για τη Λιβύη μετά τη δικτατορία. Λοιπόν, η Ευρώπη υποτιμά ένα θέμα το οποίο εμείς δεν το υποτιμούμε γιατί ξέρουμε ότι βρίσκεται στο κέντρο των προβλημάτων. Τι σημαίνει το γεγονός λοιπόν ότι έρχονται στην εξουσία κόμματα που πρόσκειται στο πολιτικό Ισλάμ. Σημαίνει ότι προφανώς ακόμα και αν είναι κόμματα τα οποία έχουν έρθει στην εξουσία δημοκρατικά μετά από δημοκρατικές εκλογές και κόμματα τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να βρίσκονται στο πολιτικό στερεώμα των χωρών τους γιατί εκπροσωπούν ένα τμήμα του πληθυσμού, είναι χώρες, είναι κόμματα τα οποία έχουν μια συντηρητική, μια αντιδραστική ιδεολογία που στρέφεται κατά των γυναικών. Δεν θα πρέπει να ψ, το θέμα αυτό και να το καλοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε σήμερα είναι η κατάσταση ισορροπίας δυνάμεων στο εσωτερικό των χωρών αυτών που είναι σε πορεία δημοκρατικοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται οι διεκδικήσεις των γυναικών αυτή τη στιγμή. Προφανώς είναι διαφορετικές οι ισορροπίες δυνάμεων από χώρα σε χώρα και οι εικόνες που είχατε της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Τινησίας, του Μαρόκου δεν είναι παντού η ίδια πραγματικότητα, δεν είναι σε ίδια κατάσταση η πρόοδος των, είναι των δικαιωμάτων των γυναικών. Θα πάρω δύο παραδείγματα μονάχα, τα οποία δίνουν το γενικό πλαίσιο. Η Τινησία είναι μια χώρα όπου η διαδικασία εκκοσμίκευσης είναι προχωρημένη, λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Τινησία είναι μια χώρα όπου το κόμμα Ενάχτα είχε δυσκολία να εξασφαλίσει ότι θα γίνουν δεκτές οι προτεραιότητές τους. Δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθεί, αλλά δεν το έχει πετύχει πλήρως. Ακόμα και αν είναι τακτική αναδίπλωση, η Τινησία μαζί με τον Λίβανο είναι οι μόνες αραβικές χώρες που δεν ισχύει η Σάρια. Η Ενάχτα λοιπόν είχε προτείνει να είναι πηγή δικαίου η Σάρια και τελικά αναγκάστηκε να ανακαλέσει μετά από μια ευρεία αντεπίθεση της κοινωνίας των πολιτών. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορέσουν να το πετύχουν με άλλους τρόπους. Αντίθετα στην Αίγυπτο το άρθρο 2 του Αιγυπτιακού συζητάγματος λέει ότι η Σαρία είναι η κύρια πηγή δικαίου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι ομοιόμορφα τα πράγματα και η ισορροπία δυνάμεων δεν είναι ακριβώς η ίδια. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχει χαθεί το παιχνίδι. Το είπατε κυρία Μπαντράν με πολύ σωστό τρόπο. Οι ίδιες οι επαναστάσει δεν έγιναν στο όνομα τη θρησκεία. Δεν έγιναν με συνθήματα αντιδραστικά ή συντηρητικά. οι επαναστάσεις στην Τίνιδα και στο Κάιρο έγιναν με το σύνθημα της αξιοπρεπίας, της δημοκρατίας, του τέλους της διαφθοράς. Το κίνημα του πολιτικού Ισλάμ, για λόγους που δεν προφταίνω τώρα να σας εξηγήσω, μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το λαϊκό κίνημα και την επαναστατική κατάσταση. Πιστεύω όμως παρόλα αυτά, και το είπαμε, ότι λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτήν την ισορροπία δυνάμεων και τον δυναμισμό της κοινωνίας των πολιτών. Και την σχετική, η σχετική ελευθερία που υπάρχει σήμερα επιτρέπει σε αυτή την κοινωνία των πολιτών να αρθρώσει τις απόψεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τώρα διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή δεν έχουν μεγάλο λόγο στο πολιτικό επίπεδο. Πολλές ε, οργανώσεις, πολλά κόμματα επενδύουν στην κοινωνία των πολιτών για να αντισταθμίσουν την απουσία του από το πολιτικό στίβο. Και έχουν αυτό το σημαντικό, αυτή τη σημαντική διεκδίκηση που είναι η, συντα... η εγγραφή στα συντάγματα των δικαιωμάτων και της ισότητας ανδρών και γυναικών και η εγγραφή στο Σύνταγμα της Αρχής της Μη Διάκρισης. Από το 2006 στο Ραμπά μια συμμαχία σε όλο το κόσμο που φέρει το όνομα Ισότητα χωρίς επιφυλάξεις. Από το 2006 λοιπόν συνενώνει διάφορες φεμινιστικές οργανώσεις στο Μαρόκο, στο, στην Τινησία. Είναι τμήμα της Διεθνούς Νομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Γυναικών από το 2006 έως το 2011. Αυτή η Περιφερειακή λοιπόν Συμμαχία έχει ζητήσει να μην υπάρχουν πια άλλες επιφυλάξεις για τη Σύμβαση ΕΝΤΕΟ. Και το κυριότερο είναι η συμπερίληψη αυτού στα συντάγματα. Δύσκολος θα είναι ο αγώνας διότι οι κοινωνίες του αραβικού κόσμου είναι διηρημένες. Υπάρχουν μεγάλο τμήμα της κοινή γνώμης που είναι συντηρητικό. Και επειδή δεν προλαβαίνω να συζητήσω την έννοια της παράδοσης θα έλεγα είναι και παραδοσιακό μεγάλο τμήμα της κοινωνίας αν και υπάρχει ένα άλλο τμήμα που είναι υπέρ προοδευτικών ιδεών και των γυναικών. Τι μπορεί να κάνει η Ένωση λοιπόν. Κάτι που δεν έκανε κατά τη διάρκεια των δικτατοριών. Να σεβαστεί τις ίδιες τις αξίες της. Όπως ξέρετε όλες οι συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ Ένωσης και διαφόρων χωρών είχαν στο άρθρο 2 το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπάθησε να επικαλεστεί αυτό το άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης για τις ελεύθερες συναλλαγές στις σχέσεις της με τις δικτατορίες του νοτίου τμήματος της Μεσογείου. Αυτό να κάνει από τώρα. Αυτό νομίζω θα βοηθούσε πολύ τις γυναίκες ε, σε αυτό το τμήμα της Μεσογείου αν θεωρούμε ότι τα γυναικεία δικαιώματα είναι και αυτά ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπεσής. Να σας υπενθυμίσω ότι στις συμφωνίες αυτές προβλέπεται σε όλες τις συμφωνίες σύνδεσης να υπάρχει μία ρήτρα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης και μια ρήτρα σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και πρόσφατα έχει εισαχθεί αυτή η ρήτρα χάρη στις προσπάθειες και την πίεση της δικής μας Επιτροπής και έχει πράγματι εισαχθεί και στις πρόσφατες συμφωνίες η τελευταία ρήτρα του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών. Όπως ελέγχθη, το βασίλειο της εξουσίας είναι το ανδρικό βασίλειο και γι' αυτό οι ηγέτες μας, ακόμα και στην Ευρώπη, έχουν άλλες προτεραιότητες. Λένε τα λόγια αυτά για τον αγώνα κατά των διακρίσεων, την ισότητα των φίλων τα δικαιώματα των γυναικών και όλα αυτά. Όλα αυτά τα ωραία λόγια τα οποία δεν υλοποιούνται όμως και δεν αποτελούν προτεραιότητες. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού και να αγωνιζόμαστε για την τροποποίηση αυτής της κατάστασης του λεχθέντος. Έχουμε την κυρία Νεντέλτσεβα και την κυρία Κουρμάη που έχουν ζητήσει το λόγο και που θέλουν να κάνουν σχόλια σε αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία λέχθηκαν από το τελευταίο πάνελ. Η κυρία Νεντέλτσεβα είναι ευρωβουλευτής και ανήκει στην ομάδα του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τις τρεις ομιλήτριες για τις εξαιρετικές τους παρεμβάσεις. Κυρία Μπεσής, με συγχωρείτε, θα αρχίσω από εσά πρώτα, που ήταν η τελευταία ομιλία. Εγώ σέβομαι πολύ το ΕΦΙΔΕΑ στην Παναγκόσμια, την Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχω πολλές φορές βασιστεί στη βοήθειά σας, αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη διαφωνία μου με αυτά που είπατε. Πρώτον δηλαδή ότι η Επιτροπή Γυναικών δεν δουλεύει σοβαρά. Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Ίσα ίσα χάρη σε εμά μπορεί να ακουστεί η φωνή των γυναικών. Δεύτερον, πιστεύω στην αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας και με ενοχλούν αυτά που είπατε ότι από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη οι γυναίκες της Βορείου Αφρικής. Εγώ είμαι υπέρ της αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών. On a parlé de la faible... Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι τόσο λίγες γυναίκες στα πολιτικά κόμματα, γιατί δεν ψηφίζουν τις άλλες γυναίκες. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι κάτι από τα θετικά συμπαράγματα που μπορούσαμε να βγάλουμε είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών που είναι προϋπόθεση αν θέλουμε να πάρουμε κανένα αποτελεσματικό μέτρο. Έχετε δίκιο, μας λείπουν τα συγκεκριμένα απτά μέτρα, όχι μόνο λόγια. Θα ήθελα τώρα να εκφράσω μερικές σκέψεις. Δικαίως λέτε ότι πολύ εύκολα αποκλείονται οι γυναίκες από τον κοινωνικό τομέα αυτό γιατί σε μια μετάβαση προς τη δημοκρατία ισχύει περισσότερο ως σημαντικότερο η πολιτική σταθερότητα. Αυτό έγινε και στη Βουλγαρία. Ενώ η ιδιαιτερότητα όλων των μεταβάσεων που γίνονται στη Βόρεια Αφρική είναι ότι είναι τριπλές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβάσεις ταυτόχρονα. Και εδώ βλέπω και εμπόδια αλλά και προκλήσεις για τις γυναίκες εμπόδια γιατί τους αποκλείουν από τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, από τη συγγραφή των κειμένων, αλλά και πρόκληση γιατί είναι μια ευκαιρία για να ενισχύσουν το ρόλο τους. Ο ρόλος των γυναικών στις δημοκρατικές μεταβάσεις φαίνεται από αυτά που είπατε και οι τρεις, ότι δηλαδή ο ρόλος των γυναικών είναι ρόλος κλειδί για τις τρεις περιόδους κάθε μετάβασης προ, κατά τη διάρκεια και μετά. Όταν μιλάμε για το πριν λοιπόν, όλες είπατε ότι πρέπει να μπορούν οι γυναίκες να συμμετέχουν στη συγγραφή βασικών κειμένων και να διαπραγματεύονται και αυτές τη μετάβαση. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση, να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους οι γυναίκες. Να ευαισθητοποιήσουμε τις ίδιες τις γυναίκες για να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για το κατά. Η πρόσβαση σε υπεύθυνε θέσει, οι λίγε γυναίκε που αναφέρθηκαν, η αντιπρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου κτλ. Πού βρίσκονται οι υπόλοιπε. Αυτές έστω και οι λίγες είναι υποδείγματα. Αλλά και οι άλλες που είναι εκτός της πολιτικής σφαίρας θέλουν να συμμετέχουν. Συχνά οι γυναίκες που καταλαμβάνουν υπεύθυνε θέσεις πάβουν να είναι αγωνιστικές. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να έχουμε το θάρρος να το πούμε. Όταν θέλουμε, όπως είπατε, μοντέρνα, σύγχρονα κείμενα, όπως είπε και η κυρία Χαντούς για το Μαρόκο, υπάρχουν ονειρεμένα κείμενα, αλλά το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν. Τι γίνεται με την εφαρμογή. Μπορούν οι γυναίκες να απευθυνθούν σε κάποιο όργανο για να ε, ζητήσουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. Γιατί μόνο έτσι θα έχουν εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη για να μπορέσουν να κάνουν μηνύσεις και για να ενοχλήσουν ακόμη περισσότερο όσους παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό και τελειώνω με κάτι άλλο για την συνεχή ευαισθητοποίηση. Πώς θα μάθουν οι νέοι ποια είναι η προβληματική της ισότητας των φύλων. Όταν βλέπουμε τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μπορούμε να ελπίζουμε και σε μια ηλικιακή αλλαγή αλλά την προετοιμάζουμε τη νέα γενιά και των ανδρών για να βλέπουν τις γυναίκες διαφορετικά. Αυτά είναι πράγματα νομίζω που μπορούμε να συνεχίσουμε να τα ζητάμε και στις οργανώσεις σας που εργάζονται υποδειγματικά πραγματικά. Αλλά στην Ένωση νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας και ειδικά στην Επιτροπή Γυναικών μαζί με τις άλλες είναι βασικό εργαλείο για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και όλους όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την πραγματική εφαρμογή. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε νομίζω, προσέχοντας βέβαια για να υπάρχει συνέπεια και διατήρηση της ιδιαιτερότητας της κάθε χώρας, γιατί συμφωνώ ότι δεν πρέπει να γίνονται υπερβολικά ευρείες γενικεύσεις όπως η Ανατολική Ευρώπη ας πούμε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση. Εγώ είμαι υπέρ της ιδιαιτερότητας της κάθε χώρας γιατί σημαίνει ότι έτσι σεβόμαστε και την ιδιαίτερη πορεία της και τότε και οι γυναίκες θα παίξουν το ρόλο τους όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νεντέλτσεβα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπεσίθ γιατί θέλει μετά να φύγει. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. για την παρεμβασή σας, αλλά νομίζω ότι ήταν ίσως ε, θέμα διατύπωσης και δεν ήταν θέμα ουσίας γιατί πιστεύω απόλυτα στην αλληλεγγύη. Πιστεύω πως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κατά τη διάρκεια της ε, δικτατορίας ε, τέθηκε σε δοκιμασία. Ήταν πολύ συχνά δύσκολο να κινηθεί η Κομισιόν, αλλά το Κοινοβούλιο πάντα υποστηρίζει τους δημοκράτες. Και αυτό θέλω να το δηλώσω. Αν στην Ευρώπη οι δημοκράτες στην Νότια Μεσόγειο βρήκαν συμμάχους ε, και η υποστήριξη ήταν στο Κοινοβούλιο. Αλλά η Κομισιόν εντάξει είναι τα κράτη, είναι πιο δύσκολο και γι' αυτό ακριβώς και η Κομισιόν θέτει σε εφαρμογή τις συνθήκες και όχι το Κοινοβούλιο. Και αν το άρθρο 2 χαροπά παραβιάστηκε καθ' όλη την περίοδο της δικτατορίας, αυτό δεν το έκανε το, Ευρωκοινο... το Ευρωκοινοβούλιο. Αντιθέτως, το Ευρωκοινοβούλιο διαρκώς ήταν, ε, ήταν... έκανε εκθέσεις για το θέμα της δημοκρατίας, για την ελευθερία. Γι' αυτό πρέπει να το αναγνωρίσαμε. Είχαμε πολύτιμη βοήθεια. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να πω και σε τόσο σύντομες ε, παρεμβάσεις δεν μπορούμε να τα πάμε, πούμε όλα. Για την Επιτροπή Γυναικών, εγώ δεν είμαι κατά, φυσικά και πρέπει να υπάρχουν απλά. ήθελα να πω ότι πολύ λίγο ενδιαφέρουν τους άντρες ε, που συχνά συμμετέχουν στις οικονομικές και στις ε, χρηματοπιστωτικές επιτροπές οικονομίας, ε, οικονομικών κτλ δεν ήθελα να πω ότι είναι άχρηστη, αλλά πολύ συχνά ενδιαφέρει μόνο τις γυναίκες. Αυτή τη διαπίστωση ήθελα να κάνω, δεν είναι μια ανάλυση, είναι μια διαπίστωση. Και έπειτα πιστεύω πως αυτό που είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί είμαι πεπισμένη και είναι και η τελευταία μου παρατήρηση, είμαι πεπισμένη πως βρισκόμαστε σε περιόδους μεταβατικές που θα διαρκέσουν πολύ. Δεν πρέπει κανείς να πιστεύει ότι, είμαστε, ότι τελειώνουν αυτές οι μεταβάσεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν φάσεις πρόοδου και επιστοδρόμησης. Αλλά ακόμα είμαστε στην οικοδόμηση της δημοκρατία κατά βάση. Και ένα τα βασικά, μια από τι βασικέ προκλήσει είναι οι γυναίκε να μπορέσουν να κατακτήσουν τη θέση του σε αυτές τι μεταβατικέ περίοδους. Και ξέρετε, το στο FIDAS, το Μάρτιο 2011, μετά από την Επανάσταση, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο στην Τίνιδα, ε, από χώρες ε, μετάβασης, ε, μετάβασης επιτυχούς και αποτυχημένης. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο από τις χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης, από χώρες που γνώρισαν μεταβατικές περιόδου, γιατί έχουμε πολλά να μάθουμε επίσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας ταξίδι και καλή τύχη. I give the floor to Zita σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα υπόθηκαν ότι οι άγγελοι και οι, οι φορείς της αλλαγής είναι συχνά οι γυναίκες. Και και συχνά αυτό παραβλέπεται και, και στην Ουγγαρία είδαμε παρά, κάτι παράλληλο με αυτό που συμβαίνει τώρα στην Αραβική Άνοιξη. Γιατί οι γυναίκε ήταν στην αρχή τη αλλαγή και μετά χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Πολύ σημαντική λοιπόν η σημερινή ακρόαση και η συζήτηση. Και θα πρέπει να την παρακολουθήσουν όλοι οι συνάδελφοι και να παρακολουθούν και τα ε, γεγονότα της εξελίξης οι σοσιαλιστές και δημοκράτες διοργάνωσαν μια διάσκεψη στη Βαρκελόνη τον περασμένο Ιούνιο ε, μια ευρωμασογειακή διάσκεψη που βέβαια δεν συζήτησε μόνο τις γυναίκες αλλά και τα θέματα των νέων γιατί η νεολαία είναι ένα πολύ, ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της επανάστασης και θα πρέπει να εισακουστεί. Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με ακτιβιστές από τη Λιβύη στις 30 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και η ομάδα μας διοργανώσαμε ένα φόρουμ με τίτλο «Αραβική Άνοιξη» και προοδευτική ατζέντα του αραβικού κόσμου. Αυτό ήταν ο τίτλος και στην Τίνιδα ε, επίσης υιοθετήσαμε μια δήλωση και εγώ ως ε, αρχηγό, ε, του οργάνωση των γυναικών του Σοσιαλιστικού Κόμματο, προσδίδα μεγάλη σημασία στην αφιέρωση ενό ολόκληρου κειμένου σε αυτή τη δήλωση για τα θέματα των γυναικών. Η συμμετοχή των γυναικών, ίσα δικαιώματα, είναι θεμελιώδη για αυτές τις αναδυόμενες δημοκρατίες ε. ο οικογενειακός κώδικας θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να εξασφαλίσει στις γυναίκες τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες και πραγματικά ήθελα να τονίσω πως η παιδεία είναι κρίσιμη. Χρειάζονται εκπαιδευμένες γυναίκες, μορφωμένες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων για να μπορέσουν οι γυναίκες να αποκτήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και να αποφασίζουν για το δικό τους μέλλον. Επιπλέον, η ε, το θέμα των φίλων θα πρέπει να μπει σε όλες τις ατζέντες σε αυτή την επιτροπή έχουμε επίσης και κάποιους άνδρες. Και συμφωνώ μαζί σα ότι αν θέλετε να γίνουν αλλαγές πρέπει οι άντρε να παρακολουθούν τα γυναικεία θέματα και αν κανείς εκπαιδεύσει τις γυναίκες σε μια κοινωνία μπορεί να εκπαιδεύσει ταυτόχρονα και τους άντρες. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε εμά και στου άντρε αλλά το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ακούσαμε επίσης τα όσα είπε η κυρία Μπαντράν για την επανάσταση, ότι οι γυναίκες παίρνουν το πιστοποιητικό τους ε, υγείας ε, επειδή καθάριζαν και τις πλατείες, είχαν τριπλό ρόλο. Και όταν μιλάμε για μοιρασιά τη εξουσία, τότε βέβαια τι ξεχνάνε τι γυναίκε. Και φυσικά το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, για παράδειγμα να υποστηρίξει τι ε, περιφέρειε, ώστε να είναι μίνιμουμ 30% γυναίκες σε οποιαδήποτε σύσταση, σε οποιοδήποτε θεσμό. Η χειραφέτηση λοιπόν και ο δημοκρατισμός θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. να εξασφαλιστεί η οικονομική αναξαρτησία και η χειραφέτηση των ε, γυναικών και των νέων. Ο Μάρκ Ταραμπέλα, ένας από τους νέους συναδέλφους μας, ε, νέος εντοσταγωγικών, διοργάνωσε μια διάσκεψη πέρυσι και εκεί παρουσιάστηκαν διάφορα παραδείγματα ε, ε, ενώσεων που βοηθούν τις γυναίκες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, μικρή επιχείρηση στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, ναι. πράγμα το οποίο δεν μπορεί να κάνει κανείς χωρίς τη συγκεκριμένη γνώση. Να τονίσω και για την ανεργία των νέων, να σας πω ότι κάναμε μια εκστρατεία, ξεκινάμε μια εκστρατεία για την ανεργία των νέων, γιατί μιλάμε για 6 εκατομμύρια νέους άνεργους. Αν πάρουμε 10 εκατομμύρια από το κοινωνικό ταμείο, μπορεί να φτιάξουμε 3 εκατομμύρια θέσεις. Και ξέρω ότι το φαινόμενο είναι παρόμοιο. Αν πάει κανείς στην Ισπανία, στην Ελλάδα, να φτάνει και στο 50% η ανεργία των νέων αλλά έχουμε παρόμοιο πρόβλημα και πιστεύω πως και η Ευρώπη ε, κάθεται πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα και θα πρέπει και εμείς να μάθουμε από αυτές τις εμπειρίες των νέων ε, χωρών και να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τις δυνατότητες μας μέσω οδηγών ή γλωσσάρια ε, για την πρόθεση των θεμάτων της ισότητας αλλά αυτό που είναι και επίση πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη την ισότητα σε όλα τα θέματα, γιατί η ισότητα δεν είναι για τις γυναίκες, είναι για την κοινωνία. Εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα η σημερινή μας συνεδρίαση. Είμαι βεβαία ότι η κυρία Κώστα θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να τα πούμε ε, ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Ζήτα. Ε, άλλη μια αίτηση από την Άννα Γκόμις, η οποία και αυτή έχει πάει σε πολλές από τις χώρες αυτές της Βόρειας Αφρικής. Και πιστεύω ότι θα τον ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική της ε, κατάθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι τα μάλα που δεν μπόρεσα να είμαι εδώ πέρα παρούσα αυτό το απόγευμα και να ακούσω από τις εμπειρίες σας. Είναι πολύ δύσκολο να οργανώσει κανείς το έργο των ευρωβουλευτών μας και αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα και ένα σεμινάριο για την Βόρεια Αφρική όπου λαμβάνει χώρα και όπου είναι παρόν ο Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Τινησίας. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, χωρίς βέβαια να έχω ακούσει τι είπατε. Θα ήθελα να σας δώσω τη δική μου εικόνα ως εισηγήτρια για τη Λιβύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από πολλές επισκέψεις που έχω κάνει στη Λιβύη, κάθε μήνα ουσιαστικά και έχοντας μιλήσει σε ακτιβιστές από την Τινησία και την Αίγυπτο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο θα μπορέσει να το βάλει η Σοφία στην έκθεσή της για να μεταλαμβατευτεί στην Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι θα πρέπει να περάσουμε από τις λέξεις, τις πράξεις αμέσως. Αμέσως σημαίνει έπρεπε να το είχαμε κάνει χθε ή και προχθές. Να βοηθήσουμε τις γυναίκες, όπως είπε η Τσίτα, να οργανώσουν τις γυναικες οπως ειπε η τσιτα να οργανωσουμε τις ικανοτητες τους να κατέβουν στι εκλογές του υποψήφιε και αφού εκλεγούν να τις βοηθήσουμε στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Το να συμμετέχουν οι γυναίκες στον πολιτικό χώρο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να εξασφαλιστεί η δημοκρατία στις χώρες αυτές, όπου και στην Ευρώπη και στην Ευρώπη δεν είμαστε τέλεια δημοκρατία, όπως ξέρετε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο τώρα και πρέπει να ασκήσουμε όλη την πίεση που μπορούμε στην υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και στη Λέδη Άστον και τις υπηρεσίες της για να μπορέσουμε σε όλες αυτές τις χώρες να έχουμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι θα αλληλεπιδράσουν με τις γυναίκες. Θα βοηθήσουν τις γυναίκες στην εξουσία, θα κινητοποιήσουν ΜΚΟ ευρωπαϊκές που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη για να εργαστούν μαζί τους για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό στίβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει χθε. Είναι κάτι που θα γίνει, πρέπει να γίνει αμέσω. Ευχαριστώ, Άννα. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τις προσκεκλημένες μας που έλαβαν το λόγο σε αυτό το πάνελ αν θα θέλαν να κάνουν κάποια σχόλια. Συγγνώμη. Πριν δώσω το λόγο στις εμπειρογνώμονες για τα τελικά της σχόλια, θα ήθελα να ζητήσω από την εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση και μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να λάβω το λόγο. Είμαι στα Ηνωμένα Έθνη τη Βρυξέλλε και εργάζομαι για τα θέματα αυτά. Είναι δύσκολα τα θέματα για την ισότητα των γυναικών. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όλε οι γυναίκε να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Στι πολιτικέ μεταλλαγέ. Οι ήδη οργανωμένε ομάδε συμφερόντων είναι πολύ ισχυρέ και ικανέ να παίρνουν εξουσία, ενώ είναι υποχρηματοδοτημένε οι οργανώσει των γυναικών και όχι σε θέση να μπορέσουν να, να επηρεάσουν την πολιτική. Mm. Είναι σαφέ ότι οι γυναίκε θα αντιμετωπίσουν σημαντικέ δυσκολίε για να εξασφαλίσουν ισότητα συμμετοχή στον πολιτικό στίβο. Πρέπει να κάνουμε ε, να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση όπου οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ε, υλοποιηθεί σε κατάληψη θέσεων εξουσίες. Ενώ η Αραβική Άνοιξη έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει ισότητα των γυναικών έχει κάνει τροτές τις ε, επιτυχίες των γυναικών στο παρελθόν. Σε πολλές χώρες όπως με την Ισία, Αιγύπτος και η Λιβύη είναι ρευστή η κατάσταση. Θα πρέπει να τονίσουμε και να συνεχίσουμε να επιμένουμε στην πολιτική των γυναικών στον πολιτικό χώρο, ώστε τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα των γυναικών να προασπιστούν και να εγγραφούν στα νέα συντάγματα. Πρέπει να έχουμε μια πραγματική αλλαγή η οποία εξασφαλίζει τα ίσα δικαιώματα όλων των πολιτών και που θα δώσει στις γυναίκες αλλά και στους άντρες την ίδια ικανότητα συμμετοχής. Αυτό το χρονικό διάστημα μετάβασης είναι σημαντικό και για τις γυναίκες και αυτούς που επιζητούν τη δημοκρατία. Πρέπει να δώσουμε και περαιτέρω δυνατότητες σε οικονομικό επίπεδο γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανοιγία των γυναικών σε όλο τον κόσμο στον αραβικό χώρο. Ξέρουμε ότι η απασχόληση των γυναικών ε, δίνει δυνατότητες στις γυναίκες και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική ισότητα συγχρόνως μαζί με άλλες ε, ε, εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τι ελευθερίε και τα δικαιώματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή του στην περιοχή αυτή, λαμβάνοντα υπόψη τι διάφορε προκλήσει που αντιμετωπίζει κάθε χώρα και τι διαφορετικέ καταστάσει που έχει κάθε χώρα. Σε αυτή τη στιγμή ιστορική αλλαγή δεν μπορούμε να αφήσουμε τι γυναίκε στο περιθώριο. Πρέπει να υπάρχει πλήρη και ίση συμμετοχή του στον πολιτικό χώρο για να εξασφαλίσουν τη δημοκρατία και την δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μονσεράτ Πρέντα. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τις ειδικέ μας προσκεκλημένες ε, για να προβούν στα τελικά του σχόλια, ξεκινώντας ε, με την κυρία Αντούσου αν το επιθυμεί. Μήπως θέλετε να κάνετε τελικά σχόλια. Όχι, ήθελα να πω τα εξής. απαντησούλες σε μερικά πράγματα που ακούστηκαν. Να αντιδράσω δηλαδή στο τι μπορούν να πούν τα κράτη, ας πούμε τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιαιτερότητες. Εγώ συμφωνώ με την συνάδελφο για το πρόβλημα της εφαρμογής όλων όσων λέμε. Πράγματι όταν ζητούσαμε αλλαγή της νομοθεσίας οι νόμοι μεν εγγυώνται τα δικαιώματα των γυναικών μπορούν να τις στηρίξουν για να εκφράσουν αιτήματα αλλά στην εφαρμογή υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει το πρόβλημα των ανθρωπίνων πόρων, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, την απόσταση των δικαστηρίων, ο αναλφαβητισμός που μειώνει την πρόσβαση στα δικαιώματα και το πρόβλημα της ίδιας της ερμηνείας των κειμένων γιατί οι δικαστές ερμηνεία κάνουν όχι μαθηματική εφαρμογή, ερμηνεία. Στο Μαρόκο έγινε ένα βηματάκι ως προς την εκπαίδευση των δικαστών. Υπήρξε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των δικαστών και μία γνωστή φεμινίστρια συμμετείχε Υπάρχουν λοιπόν, έγιναν πράγματα τώρα. Όντως υπάρχει το άλλο πρόβλημα, το άλλο. Κατά πόσον οι πολίτες δέχονται ή όχι τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Πολλοί λένε ότι δεν έπρεπε να μεταρρυθμιστεί ο οικογενειακός κώδικς. Άλλοι λένε ότι το γυναικείο κίνημα ζητάει κυρίως την ισότητα στην κληρονομία και αυτή είναι αντίθετη. Είναι δύσκολο να δουλέψει κανείς με τέτοιο κλίμα, αλλά το, το κατορθώνουμε παρόλα αυτά. Μέχρι τώρα διστάσαμε να πούμε κάτι για την κληρονομία διότι κάθε φορά εξετάζουμε αν το επιτρέπει αυτό το κοινωνικό κλίμα. Για τους εκλογικούς καταλόγους τώρα, για να μην κάνουν οι άλλες χώρες το ίδιο λάθος. Εμείς δεχτήκαμε τον εκλογικό κατάλογο που ε, προέβλεπε 36 έδρες για γυναίκες. Είπαμε δεν πειράζει, μια αρχή είναι. Μετά θα αυξηθεί η ποσόστοση, αλλά τελικά μέχρι τώρα δεν αυξήθηκε. Και όταν ζητούμε από τα κόμματα στα ψηφοδέλτια τους να συμπεριλαμβάνουν γυναίκες και επικεφαλής του ψηφοδελτίου λένε όχι αυτές έχουν χωριστό ψηφοδέλτιο και τελικά παραμένουμε στον αριθμό εκείνων των 30 γυναικών. Επίσης για τις μελλοντικές γυναίκες τα Ισλαμιστικά κόμματα τελικά προτείνουν περισσότερες γυναίκες. Μπαίνουν στη Βουλή λοιπόν οι γυναίκες, θα αλλάξουν όμως την κατάστασή τους. Θα ζητήσουν ισότητα. Τέλος, για σας, για σας, την ιδιαιτερότητα. Κάθε φορά που μερικοί συζητούν με τους ηθήνοντες για τα γυναικεία δικαιώματα, τους λένε αυτό είναι θέμα ιδιαιτερότητας. Όχι, δεν είναι ιδιαιτερότητας, είναι ανθρώπινα δικαιώματα αυτά. Είναι παθολικά παγκόσμια. η θρησκεία είναι θρησκεία. Δεν μπορεί να επικαλεστεί ιδιαιτερότητα. Είναι μια θρησκεία. Το αίτημα να μην βασίζεται η νομοθεσία στη θρησκεία δεν το δέχτηκαν πάντως. Αυτά. Ναι, αλλά να σεβαστούμε και τα δικαιώματα των ερμηνευτριών ε, δεν πρέπει να ξεπερνάμε το χρόνο μας λοιπόν. Έχετε, θέλετε να μιλήσετε. Ορίστε. Μόνο να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Κώστας τι θα κάνουμε αφού μας έχουν βάλει στον τοίχο με τον Σαφέκ και τον Μούρση. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα πάμε να ψηφίσουμε αλλά όχι τον έναν ή τον άλλον οργανώνουμε γραπτός ότι δεν τους θέλουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Θα βάλουμε άκυρο ψηφοδέλτιο, θα γράψουμε πάνω όχι. Και όταν εκλεγεί ο Σαουφίκ, γιατί θα εκλεγεί, διότι ο στρατός θα τον φέρει με τελείως μη δημοκρατικές διαδικασίες, όταν έρθει στην εξουσία λοιπόν θα ξέρει ότι δεν είναι και τόσο δημοφιλής θα ξέρει ότι υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν τον θέλουν και κατά την τετραετή θητεία του δεν θα μπορέσει να κάνει ό,τι θέλει. Δεύτερον, ευχαριστώ την Κομισιόν που είπε ότι φέρνει περισσότερους πόρους στη Βόρεια Αφρική. Ελπίζω ότι δεν δίνει απλώς λεφτά αλλά θα παίξει το ρόλο εταίρου, θα έρθει επί τόπου, θα συνεννοηθεί μαζί μας, θα μας κάνει capacity building που λένε. Θέλουμε ενεργή αλληλεγγύη, πραγματική εταιρική σχέση. Τρίτον, είπε κάποιος ότι πρέπει να σταματήσουμε πια τα λόγια. Εμεί τα έχουμε σταματήσει, δεν περιοριζόμαστε στα λόγια οργανωνόμαστε για δράση και επίσης καταλαβαίνουμε ότι έχουμε προβλήματα και μεταξύ μας οι γυναίκες καμιά φορά όταν γίνονται ηγέτησες δεν υποστηρίζουν τις άλλες γυναίκες. Προσπαθούμε λοιπόν να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό όχι μόνο εμείς αλλά όλη η κοινωνία των πολιτών με τις διασυνδέσεις της με συνδικάτα να παίζει ρόλο αλληλεγγύης πράγματι. Και τώρα θα καλέσω την Επιτροπή να, να πάρει το λόγο για να κάνει τα τελευταία της σχόλια. Okay. Uh, yes, please. Je, je parlais de la Libye